Okay. Uh, just... Αρχίζουμε λοιπόν. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έγκριση τη ημερήσιας διάταξη είναι το πρώτο μα θέμα. Αν δεν έχετε διαφωνίε και αντιρρήσει, εγκρίνεται. Θα ήθελα... Mm, Να σας επιστήσω την ε, προσοχή στο εξή. Δανικά, ε, κροατικά και ιρλανδικά δεν έχουμε σήμερα. Αύριο ψηφίζουμε στις 11.40 και παρακαλώ να έχετε μαζί σας τις ε, κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 30 Μαρτίου 2017, 26 Σεπτεμβρίου 2016 και 11 και 12 Ιουλίου του 2016. Αν δεν διαφωνείτε, εγκρίνονται. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την εξωτερική διάσταση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης και έχει σχέση με την ε, διακήρυξη της Μάλτας ε, του Φεβρουαρίου 2017, όπου το Συμβούλιο αποφάσισε να ε, αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τη Λιβύη. Καθώς η Λιβύη είναι μια βασική χώρα ε, προέλευσης αλλά και διέλευσης μεταναυστών. οι οποίοι έρχονται μέσα από την κεντρική Μεσογειακή Πάνω από 180.000 είναι οι ιδιαίτερα στην Ιταλία το 2016 και ε, αριθμός ρεκόρ πνιγμών σημειώθηκε στη ε, Μεσόγειο αρχές του έτους στην προσπάθεια των προσφύγων να διασχίσουν τη θάλασσα. Συνεπώς, μετά από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, όπου παρατηρήθηκε μείωση της ε, άφηξης ε, των αφήξεων καλύτερα από την Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνονται αφήξεις από τη Λιβύη. Μετά την διακήρυξη της Μάλτας, ε, αυτό σημαίνει ότι είναι προτεραιότητα της Ένωσης να σταθεροποιηθεί η Λιβύη. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τις αρχές να ανακτήσουν την κυριαρχία και τον έλεγχο των χωρών, της χώρας μάλλον και των υδάτων. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα που αναφέρονται στη διακήρυξη μάθηση. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε δύο από αυτά. Την υποστήριξη και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων στην ε, Λιβύη, ιδιαίτερα στις παράκτες περιοχές. Και επίσης ε, βοήθεια για να βελτιωθεί η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και να ενισχυθεί η ικανότητα της ε, Λιβύης ε, να υποδέχεται πρόσφυγες. Επίσης, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι σωστές εγκαταστάσεις και συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας για τους μετανάστες στη Λιβύη σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση. Έχουμε συναδέλφου από την Επιτροπή Εξωτερικών προσκεκλημένους να συμμετέχουν στην παρούσα συνεδρίαση. Αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εργασιών μας. Την περασμένη εβδομάδα ε, μέλη της Επιτροπής μας επισκέφθηκαν την Ιταλία για να διαπιστώσουν επιτόπου τις βελτιώσεις και τις εξελίξεις σχετικά με την οδό αυτή τη μεταναστευτική της Κεντρικής Μεσογείου. Συναντηθήκαμε με το Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοφυλακή ε, για να δούμε πώς υποστηρίζουν την καταπολέμηση της διακίνησης ε, ανθρώπων. Άρα έχει απολύτως νόημα να κοιτάξουμε και τι γίνεται στη Λιβύη σε συνεργασία με τους συναδέλφους της ΑΦΕΤ. Ε, καταρχάς θα ακούσουμε μια παρουσίαση των γιατρών χωρίς ε, ε σύνορα και ε, σε σχέση με την ε, κατάσταση των κέντρων κράτησης στην Λιβύη και τους συντονιστές που οι συντονιστέ μα το ζήτησαν αυτό. Και μετά θα ακούσουμε δύο εκπροσώπους, ένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα από την Υπηρεσία Εξωτερική Ε, είναι τιμή μου να υποδέχουμε την κυρία Αν Μαρή Λούφ, ε, που είναι η διαχείριση του προγράμματος για τη Λιβύη, και την κυρία Ινα Βάσκετ, ε, πρόσωπο της ε, Οργάνωση Γιατρών χωρί Σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σα δώσω το λόγο κυρία ε, Λούφ, για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω. Εργάζομαι για τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Από το 2015 έχουμε δύο σκάφη για τους σκοπούς της διάσωσης στη Μεσόγειο για να περισσότερους αυτού αυτούς που προσπαθούν να φύγουν. Έχουμε ακούσει φοβερές ε, ιστορίες για το τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι στην Λιβύη. Αυτό μας όθησε να μεταβούμε επί τόπου και να δρομολογήσουμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους μετανάστες και να, προλάβουμε, να τους προλάβουμε πριν να αποπειραθούν να διασχίσουν την Μεσόγειο. Είμαστε λοιπόν σε μοναδική θα θέση, έχουμε ειδική γνώση των εξελίξεων στην ε, Λιβύη, είμαστε οι μόνοι που έχουν παρουσία στην περιοχή. Ε, υπάρχουν και άλλοι βεβαίως οργανισμοί, αλλά με προσωπικό που αποτελείται αποκλειστικά από Λίβιους, σε αντίθεση με εμά δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρουσία σε περίπου 10 κέντρα στην Τρίπολη και τη Μισράτα. Μιλάμε με κρατουμένους ε, σε καθημερινή βάση ως εκ τούτου. Οπότε είμαι εδώ για να καταθέσω την εμπειρία μας και για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις σχετικές αποφάσεις της. Ο δρόμος της μετανάστευσης, όπως βλέπετε εδώ, οδηγεί, όπως όλοι οι δρόμοι, όχι στη Ρώμη προκειμένου, αλλά στην Τρίπολη. Για όσους θέλουν ε, να φύγουν από τη χώρα, η Τρίπολη είναι η υποχρεωτικό σημείο διέλευσης. Επισκεφτόμαστε λοιπόν καθημερινά κρατουμένους, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά ε, έχουν και πολλά κοινά στοιχεία και ένα από αυτά είναι ο εξαιρετικά περιορισμένος χώρος που τους διατίθεται. Πρόκειται για ακραία συμφόρηση. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν σε χώρους που δεν είναι για ανθρώπους, είναι πρώην αποθήκες. Απλώς προσθέθηκαν κάποιες ε, τουαλέτες. Στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι τυχεροί άνθρωποι. Και σε αυτές τις εγκαταστάσεις βρίσκονται συνωστισμένοι αυτοί οι άνθρωποι πριν από ένα χρόνο όταν ξεκινήσαμε συνειδητοποίησαμε ότι σε πολλέ περιπτώσει αντιστοιχούσε λιγότερο από μισό τετραγωνικό μέτρο σε κάθε κρατούμενο. Κατανοείται ότι οι άνθρωποι αυτοί ίσα ίσα που κάθονται με μαζεμένα τα πόδια δεν μπορούν καν να ξαπλώσουν. Μιλάμε για ακραία συμφόρηση. Δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχει εξαιρισμό. Οι κρατούμενοι δεν έχουν την δυνατότητα να βγουν, να προαυλιστούν ε, παραμένουν περιορισμένοι σε αυτόν τον εσωτερικό χώρο για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κέντρα αυτά λέγονται ε, κέντρα κράτησης, ε, κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, αλλά πρόκειται εν τέλει για αποθήκες ανθρώπων. Αυτές που βλέπετε εδώ είναι οι συνθήκες σε όλα τα κέντρα κράτησης. Ε, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει όταν επί μέρες και εβδομάδες άνθρωποι βρίσκονται συνοστισμένοι σε αυτόν τον χώρο. Πρόκειται για ιδανικό πεδίο διάδοση ε, ασθενειών και μολύνσεων. Μιλάμε με αυτού του ανθρώπου, παρέχουμε ιατρική φροντίδα. Οι άνθρωποι αυτοί μα πλησιάζουν, πολλοί παραπονούνται για ασθένειε άλλοι μα λένε ότι είναι εκεί επί μήνε. Ε, το 11 μήνε, για παράδειγμα το ακούμε πολλέ φορέ. δεν ξέρουν γιατί είναι εκεί, γιατί κρατούνται. Κάποιοι μάλιστα διαθέτουν και έγκυρες θεωρήσεις, μπορούν δηλαδή να ζήσουν νόμιμα στην Λιβύη. Τους μάζεψαν όμως, ε, τους κατέγραψαν ε, μέσω της ΥΠΑ του ΙΕ για τους πρόσφυγες και παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να κρατούνται σε αυτά τα κέντρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα τους κρατήσουν ακόμη. Δεν έχουν μέσα να μάθουν τι πρόκειται να τους συμβεί, να επηρεάσουν την κατάστασή τους. Βρίσκονται λοιπόν σε μια κατάσταση για την οποία δεν έχουν ιδέα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα λοιπόν. Η οικονομία της Λιβύης εξαρτάται, ή μάλλον να, ξ, να ξαναρχίσω, η εμπλοκή με τους πρόσφυγες έχει πολύ χρήμα, έτσι, για να το θέσω πολύ απλά. Αυτό αποτελεί μεγάλη πηγή ανησυχίας, διότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους, όχι για εμπορεύματα, αλλά δυστυχώς έτσι τους μεταχειρίζονται, τους πουλάνε, τους αγοράζουν. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει εμέσως έναν πρόσφυγα, να τον πάρει σπίτι του, πληρώνοντας κάποια λεφτά. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της καταναγκαστικής εργασίας ή της αναγκαστικής πορνείας στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, πρόκειται σχεδόν για συνθήκες σύγχρονου δουλεμπορίου. Η τύχη εδώ στο συγκεκριμένο οίκημα ε, είναι υγρή, διότι οι κρατουμένοι ουρούν δεν έχουν ε, πρόσβαση στην τουαλέτα και αναγκαστικά κάνουν τι ανάγκε του στον χώρο αυτών. Επίση, κρύο και στην Τρίπολη και στη Μισράτα. Δεν υπάρχει φυσικά κεντρική θέρμανση, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία θέρμανση. Οι άνθρωποι αυτοί προστατεύονται με κάποιες κουβέρτες τυποδό, αλλά στο κρύο και οι κουβέρτες αυτές φυσικά δεν αρκούν. Όπως βλέπετε αυτή είναι η κατάσταση. Και οι κουβέρτες είναι πάλι ιδανικό πεδίο ε, διαβίωσης ε, για ψήρε, ψηλού κλπ. Επίσης κρατούνται γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες κρατούνται ξεχωριστά από τους άντρες, έχουν ε, ευτυχώς έτσι λίγο περισσότερο χώρο στη διάθεσή τους, αλλά και πάλι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί. Επίσης ε, είδαμε πολλά παιδιά που μένουν με τις μανάδες τους, ε, έχουμε και νεογέννητα και πολλά παιδιά κάτω των πέντε. Κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι καλό για την ψυχική ή σωματική τους υγεία. Πρόκειται για κρατουμένους οι έγκυε, οι γυναίκες και τα παιδιά δεν θα πρέπει να κρατούνται. Αυτή είναι η πάγια θέση μας. Παρ' όλα αυτά ήταν δύσκολο να προωθήσουμε το θέμα αυτό με την κυβέρνηση της Λιβύης βάσει της σύμβασης του 1951. Μια άλλη ευπαθής ομάδα που παρατηρούμε είναι, είναι τα ασυνόδευτε, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, χωρίς και μόνα οι γονείς. Υπάρχουν αρκετοί και τους βλέπουμε και στα σκάφη τα οποία διασώζουμε στην Μεσόγειο, στη θάλασσα. Άλλη μια λοιπόν ευάλωτη ομάδα η οποία ε, επιδέχεται εκμετάλλευση. Ήδρευση, αποχέτευση, υγιεινή. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ε, οι συνθήκες δεν είναι καλές. Να το θέσω επίκως. δεν υπάρχουν τουαλέτες, πολλές φορές είναι εκτός των κοιλιών κράτησης, των χώρων κράτησης, πολλές φορές δεν υπάρχει πρόσβαση. Τώρα η ποιότητα του νερού, το νερό το οποίο υποτίθεται είναι πόσιμο νερό, είναι συνήθως κακής ποιότητας και δεν υπάρχει πρόσβαση σε σαπούνι ή άλλα καθαριστικά. Οι χώροι δεν καθαρίζονται, οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να πλύνουν τα ρούχα τους ή να κάνουν ε, ντους. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να διανεμηθούν τέτοια είδη καθαρισμού και τομικής υγιεινής από εμάς και από άλλους οργανισμούς. Είχαμε όμως αναφορές ότι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και όταν τα ίδια αυτά διατίθενται, δυστυχώς κατάσχονται. Υπό αυτά συνθήκας μπορείτε να φανταστείτε ότι οι συνθήκες υγιεινής και υγεία είναι κακές. Αυτό επηρεάζει την σωματική και πνευματική ψυχική υγεία αυτών των ανθρώπων, ε, έχουμε θανάτους. Στην εικόνα αυτή εδώ βλέπετε δύο ενηλίκους, οι οποίοι είναι θύματα υποσυτισμού. Εδώ μιλάμε τώρα για, για ενηλίκους. Ε, είναι δύσκολο να δει κανείς ενηλίκους αυτήν την κατάσταση. Έχουμε πολλά κρούσματα λοιπόν υποσχετισμό, αλλά σπάνια τα βλέπουμε σε ενηλίκους. Εδώ ε, υπογραμμίζω για μια φορά ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε εδώ είναι ενήλικοι, είναι πιο σε σε σε ασθένειες και φυσικά σε μετάδοση ασθενειών. Σε αυτούς που είναι σε χειρότερη κατάσταση, καμιά φορά καταφέρνουμε να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομείο. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν άλλα προβλήματα, τα προβλήματα του συστήματος υγείας της Λιβύης, διότι από το 2011 Σύμφωνα με μελέτες, οι συνθήκες του συστήματος υγείας στην Λιβύη έχουν επιδεινωθεί σοβαρά. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη πόρων, άρα λοιπόν και να μεταφέρουμε κάποιον σε νοσοκομείο, σε πολύ κακή κατάσταση, δεν θα λάβει την περίθαλψη που του χρειάζεται. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί υποσυτίζονται, το ανέφερα όμως αυτό προηγουμένως, αλλά το υπογραμμίζω για άλλη μια φορά γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ε, άλλοι κρατούνται σε απίστευτες ε, συνθήκες, βασικά αφήνουν να πεθάνουν ε, εξαιτία της διάρειας, της, του υποσυτισμού, της έλλειψης νερού. Εδώ βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος αφέθηκε να πεθάνει σε, ένα, σε μια τουαλέτα μετά από τρεις ημέρες. Παρατηρούμε πολλές ασθένειες δερματικές, ψωρίαση, δερματίδες. Επίσης έχουμε εγκάβματα αυτού του τύπου. Πολλές φορές η επαφή, μακρόχρονη επαφή με το νερό της θάλασσας προκαλεί εγκάματα αυτού του τύπου ε, ε, στην περίπτωση ειδικά που κάποιος δεν ε, τη χάνει άμεσης περίθαλψης. Επίσης, είχαμε θέματα, θέματα ξυλοδαρμού. Τα βράδια κάποιοι μας κατήγγειλαν ότι χρησιμοποιούνται ραβδιά με τα οποία τους δέρνουν. Κάποιοι άλλοι βασανίστηκαν σε αυτά τα κέντρα. Οι γιατροί έχουν τεκμηριώσει περιπτώσεις ακραίας βίας και ακούσαμε πολλές μαρτυρίες αυτού του τύπου. Πολλοί κατήγγυλαν τέτοιου είδους περιστατικά ε, σοβαρής κακομεταχείρισης και άσκησης βίας. Τόσο κατά ενηλίκων όσο και ανηλίκων. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες από τέτοιου είδους κρούσματα. Νομίζω ότι έχετε αρκετά στοιχεία για να σχηματίσετε μια εικόνα, η κατάσταση είναι πολύ κακή. Το βασικό μήνυμα το οποίο θα ήθελα να στείλω, γιατί ξέρω ότι έχω και περιορισμένο χρόνο, είναι ότι δυστυχώς ε, το εμπόριο των ε, μεταναστών έχει πολύ χρήμα. Νομίζω ότι αν ρίξουμε περισσότερα χρήματα στο σύστημα δεν θα τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους βοηθάμε έτσι, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ενώ το ζητούμενο είναι ακριβώς το αντίθετο. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσή του. Η λύση δεν βρίσκεται στη Λιβύη. Η Λιβύη είναι το πρόβλημα και αυτό θέλω να τονίσω και να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Αυτά προς το παρόν τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βάσκε. έχει το λόγο. Κατά την ε, παρέμβαση της Αν Μαρή της ε, συναδέλφου και μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του ζητήματος μέσα στα πλαίσια της ε, χρηματοδότησης για τη Λιβύη και τη Βόρειο Αφρική. Δηλαδή πώς ε, μπορέσαμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα προγράμματα πλήρως και αμερόληπτα. Και πόσο, κατά πόσο υπάρχει ενημέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων για την εποπτεία και την προστασία και την παραπομπή αυτών των ζητημάτων και αυτό αφορά και την μετεγκατάσταση. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν από τη Λιβύη, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για μετεγκατάσταση. Και θα ήταν σκόπιμο να μας πείτε κατά πόσο υπάρχει επίπτωση και από την διαδικασία εκπαίδευσης της ακτοφυλακής. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 7 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Λιβύη θεωρείται μία ε, μεικτή κατάσταση μετανάστευσης. Δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες και επειδή υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για την προστασία και των μετανοστών και των προσφύγων και να υπάρχει ε, πραγματική προστασία. Αυτός είναι ο απότερος στόχος και της διεθνούς κοινότητας. Ο δικός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές πρωτίστως, γιατί ξέρετε ότι η οδός της κεντρικής Μεσογείου είναι πολύ επικίνδυνη. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ε, καιρικές συνθήκες. Τουλάχιστον 4.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2016 και γι' αυτό θα πρέπει να διασώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω σε ε, βάρκες υπερφορτωμένες που δεν, έχουν αυτό τον, δεν υπηρετούν αυτό τον σκοπό και θα ε, αναφερθώ και στο θέμα της εκπαίδευσης των ακτοφυλάκων. Γιατί το εγχείρημα Σοφία είναι να κατακαιρματίσουμε αυτό το δίκτυο των διακινητών, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς ε, απόλυτα σε όλα τα επίπεδα, που δυστυχώς ε, έχει, ε, παρουσιάζει αυξημένους αριθμούς στη Λιβύη. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να βελτιώσουμε και τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσω. ο εκπρόσωπός σας στη Λιβύη, συναντήθηκα με τον εκπρόσωπό σας στη Λιβύη στην Τίνιδα μερικές εβδομάδες πριν. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους μετανάστες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επαναπατριστούν και να ενσωματωθούν στις χώρες προέλευσης. Και όπως ξέρετε, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θέλει να επαναπατρίσει 15.000, αλλά αυτή είναι μία μεγάλη πρόκληση. Επίσης, θα θέλαμε να προβάλλουμε εναλλακτικέ σε σχέση με τα κέντρα κράτησης, έτσι ώστε να υπάρχουν ανοιχτά κέντρα όπου να χορηγείται βοήθεια στους πλέον ευάλωτους. Επίσης έχει σημασία να υποστηρίξουμε τη σταθερότητα των τοπικών κοινωνιών, εκεί όπου διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η πλειοψηφία μένει σε αυτούς τους καταβλισμούς, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός ζει στην, και χρησιμοποιεί τις κοινωνικές δομές της ε, τοπικής κοινωνίας. Αυτό αφορά και τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες και ε, εκείνους οι οποίοι ε, είναι απάτριδες. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε ποιοι είναι αυτοί που ε, διακινούνται, ίσως φτάνει και το ένα εκατομμύριο στη Λιβύη. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν ήρθε στη Λιβύη για να διανύσει τη θάλασσα και να φτάσει στην Ευρώπη. Δηλαδή μεταβαίνανε στη Λιβύη αρχικά για να εργαστούν. Τώρα πια δεν υπάρχει για πολλή εργασία και βρίσκονται σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Μιλάμε λοιπόν για προστασία και σταθεροποίηση. Αυτό είναι ο απότερος στόχος με τον προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων που εγκρίθηκε στις 12 Απριλίου. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά το Ταμείο ε, Χρηματοδότησης της Βορείου Αφρικής. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Μιλάμε συνολικά για 200 εκατομμύρια. Και θα γίνει μια συνάντηση στη Μάλτα σε σχέση με την χρησιμοποίηση αυτής της χρηματοδότησης από αυτό το καταπίστευμα. Και η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης καθώς και ο ύπατος εκπρόσωπος η UNICEF και η GIZ, η γερμανική, ο γερμανικός αυτός ο οργανισμός, θα συμπράξουν. Τώρα βρισκόμαστε σε φάση υπογραφής των συμβάσεων μέχρι τα μέσα τέλη Μαΐου, για να κινηθούμε αρκετά γρήγορα. Θέλουμε λοιπόν να διαχειριστούμε καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα και αυτό αφορά την κατάρτιση των αρχών και της ακτοφυλακής έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την ε, λαθρεμπορία και την παράνομη διακίνηση, αλλά νόμιμα έτσι ώστε να μεταχειριζόμαστε τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες κατά το σωστό τρόπο. Υπάρχει και ένα νομικό χάσμα, γιατί η Λιβύη δεν συμμετέχει στη Σύμβαση της Γενέβης. Τώρα για να απαντήσω για την κατάρτιση της ακτοφυλακής της Λιβύης που άρχισε πέρσι τον Οκτώβριο. Έχουμε ε, προβεί στην εκπαίδευση των πρώτων ας πούμε ε, παρτίδων και στην ουσία μιλάμε για δύο ακτοφυλακές. Η μία ε, συνεργάζεται με το Υπουργείο Εστερικών και η άλλη με το Υπουργείο Άμυνας. Και αύριο θα μεταβούν εδώ για να μας μιλήσουν για τις ανάγκες μας. Και η ΑΕΔ θα συντονίσει αυτές τις δραστηριότητες μαζί με άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν, έτσι ώστε η βοήθεια που θα χορηγήσουμε να χορηθεί σωστά να υπάρχει σωστή δαπάνη των χρημάτων. Βεβαίω και το θέμα της πρόσβασης είναι πολύ σοβαρό, γιατί δυστυχώς και οι δικοί μας άνθρωποι που βρίσκονται στην Τίνιδα δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά αυτά τα χρήματα. Βεβαίως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα μεταβεί στη Λιβύη με την βοήθεια της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είμαστε σε θέση όμως να λάβουμε μια απόφαση και να αποστείλουμε το προσωπικό στη Λιβύη. Αλλά είμαστε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ιδιαίτερα τον κύριο Κόμπλε που είναι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στην ε, Λιβύη, στην Τίνιδα. Δεν μας απασχολεί η Λιβύη μόνο από πλευράς μετανάστευσης, θα αφήσω τον συνάδελφο να το αναπτύξει, αλλά θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση της μετανάστευσης στη Λιβύη κατά κάποιο τρόπο και αυτό είναι και η μεγάλη μας προτεραιότητα για τους επερχόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Παντηρόλη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε η κατάσταση στη Λιβύη δεν βελτιώνεται. Επιδεινώνεται η πολιτική κρίση και επίσης αυξάνεται η ανασφάλεια αλλά και οι εντάσεις μεταξύ του Λιβυκού εθνικού στρατού όπου ηγείται ο ε, στρατηγός Χάφτα και ε, των ε, ανταρτών στην Μισράτα. Ο μακροχρόνιος στόχος μας, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να σταθεροποιηθεί ένα δημοκρατικό κράτος σε ευημερία και ασφάλεια. Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Αυτό σημαίνει πρόθεση της δημοκρατίας με ένα σύνταγμα χωρίς αποκλεισμούς. Κατακτίζεται το σύνταγμα αυτό το καιρό. Έχει σημειωθεί βέβαια περιορισμένη πρόοδος, η οποία μας χαροποιεί μεν, αλλά απομένει ακόμα πολλοί δρόμο, Και θα πρέπει επίσης να οικοδομηθούν ε, γεροί θεσμοί με διαφάνεια, με κοινωνία των πολιτών και ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που από τη Λιβύη. Τώρα λοιπόν έχουμε τέσσερις βασικές γραμμές δράσης για τη σταθεροποίηση της Λιβύης. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα εξής. Πιο ενεργό συμμετοχή ε, στην υποβοήθηση της πολιτικής ε, διαδικασίας. Υποστηρίζουμε τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2015 υποστηρίζουμε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης και προσπαθούμε να φέρουμε στο ίδιο διαπραγματευτικό τραπέζι όλους τους ενεχομένους. Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη και με ε, τα γειτονικά κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς που ε, μεσολαβούν. Στις 18 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ ε, δημιούργησαν ένα νέο ε, διεθνές σχήμα για να οθήσει όλους τους ενεχομένους στη Λιβύη να συνεργαστούν στην ε, Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Όπως είπε και ο προλαλής σας, δεν μας απασχολεί μόνο η μετανάστευση. Πριν σας εξηγήσω ότι γενικότερη μας προσέγγιση στη μετανάστευση Λιβύη έχει σημασία να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 120 εκατομμύρια στα πλαίσια της διμερούς ε, ε, παροχής βοήθειας για την κοινωνία των πολιτών, την ε, δημοκρατική διακυβέρνηση, την υγεία, την παιδεία, την προστασία, την μετανάστευση, την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας και επίσης βοήθεια προς όλους όσους έχουν πληγεί από την ένοπλη σύραξη, εξωτερικά εκτοπισμένους, ε, επαναπατριζόμενους κλπ. Ε, όπως σας είπα προηγουμένως, ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την πολιτική λύση ε, στην κρίση της Λιβύης, ταυτόχρονα όμως να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα της μετανάστευσης μαζί με τους Λιβύους, ε, με προστασία των προσφύγων και καταπολέμηση των διακινητών και των δικτύων. Αυτό είναι κοινό μας στόχος και να σώζουμε τις ζωές ε, των ανθρώπων και να προωθούμε την ασφάλεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα. Έχουμε λοιπόν μια συνολική προσέγγιση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς τη Λιβύη και δια της Λιβύης. Αυτό σημαίνει συνεργασία με τις αρχές. Ε, ο κύριος Παπαύσκη εξήγησε ποια είναι η βασική μας δράση ε, που συνεχίζεται και τι προβλέπεται ε, στην συνεργασία μας με τον ΟΙΑ και την υπατιαρμοστία για τα κέντρα κράτησης και πώς βοηθούμε γενικότερα όλους όσοι πλήττονται από το θέμα αυτό αλλά επίσης συνεργαζόμαστε με τους νότιους γείτονες της Λιβύης, γιατί αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, να έρχονται όλο και περισσότεροι ε, και να κατευθύνονται προς τη Λιβύη. Προσπαθούμε λοιπόν να εντείνουμε, να αυξήσουμε τη συνεργασία μας με τους νότιους γείτονες και να ε, ενισχύσουμε την συνεργασία της ίδιας της Λιβύης με τους γείτονές της για να υπάρχει περισσότερος έλεγχος στα νότια σύνορα. Επιπλέον, καταρτίζουμε και βοηθούμε γενικότερα την ακτοφυλακή της Λιβύης, όπως είπε ο κ. Ποπόφσκι, με την ε, ε, επιχείρηση Υπόκαμος και την επιχείρηση Σόφια. Αυτό αφορά γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ε, μεταναστών. Ε, και την ε, διάλυση των ε, δικτύων των διακινητών έτσι ώστε και τα χωρικά ύδατα της Λιβύης να είναι πιο ασφαλή. Και τέλος συνεργαζόμαστε πάλι με τις Λιβυκές αρχές και πάλι θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και να ενθυμίσετε ότι δεν ελέγχουν όλη την επικράτεια οι αρχές. Προσπαθούμε και ε, για μια ε, συνεργασία ε, πολιτικό επίπεδο στη δικαιοσύνη και την αστυνομία. Η δική μας αντιπροσωπεία καθημερινά προσπαθεί να συνεργάζεται με τις λιβικές αρχές και να τους υπενθυμίσει ότι πρέπει να βελτιωθούν η κατάσταση κράτης και οι συνθήκες κράτησης των μεταναστών και των προσφύγων. Όλα αυτά βέβαια γράφονται σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο επιτόπου. Ασφάλεια δεν υπάρχει. Κυβέρνηση μία δεν υπάρχει που να ελέγχει όλη την επικράτεια της χώρας και δεν υπάρχει και πρόσβαση ε, για την παροχή βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς και προσωπικό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Not very Όχι πολύ ευχάριστα όλα αυτά, ούτε αισιόδοξα. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Και τώρα ο λόγος πρώτον στους συντονιστές της Επιτροπής μας από το ΕΛΚ. Ρομπέρτα Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ για τις σκέψεις αυτές, τις προτάσεις που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόμοιες συζητήσει βεβαίω γίνονται και αλλού. Τώρα, στην Μεσόγειο και στη Λιβύη γίνονται πράγματα που μα επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε από τη Μάλτα, από μια χώρα πολύ κοντά σε μια τραυματισμένη χώρα που περνάει δύσκολα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αμέσως. Το μόνο που δεν επιτρέπεται να κάνουμε είναι να αφήσουμε την Λιβύη να καταρρεύσει και να πέσει στα, στα χέρια του Ισλαμικού κράτου ή άλλων συνεργατών τους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν μεγαλύτερο έλεγχο τη χώρα από τους Ισλαμιστέ. Εμεί ανέκαθεν υπεραμεινόμεθα μια πιο δραστική στάση. Ε, αυτό το μήνυμα στέλνουμε και στην Κομισιόν, πρέπει το θέμα αυτό να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα. Και εμεί όμω μπορούμε να διευκολύνουμε τι συνομιλίε μεταξύ των διαφορών φατριών στη Λιβύη. Και μιλώ για φατρίε γιατί έχω συμπατριώτε μου που πηγαίνουν συχνά στη Λιβύη, τη γνωρίζουν και μου λένε όλοι ότι πρέπει ό,τι να κάνουμε το κάνουμε σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ λύσει Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει ε, από τους Λιβύους μέσω των Λιβύων. Αν θέλουμε δηλαδή να προχωρήσουμε πρέπει οι Λίβοι να εμπλακούν αμέσω. Και ας κάνουμε βεβαίω ότι μπορούμε για να υπογραφεί σύντομα μια συμφωνία. Αυτό δεν θα γίνει εν μια νύχτη. Τώρα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνεχίζουν να συζητούν, ε, χρήματα δίνονται, αλλά δεν είναι εκεί η λύση. Υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά προβλήματα. Θα έλεγα και θα πρότεινα το Συμβούλιο, οι προτάσεις της Κομισιόν και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να είναι πιο απαιτητικά στις προσπαθίες τους ε, να φτάσουμε έστω και ακόμη και σε εγκατάσταση ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή για να προστατεύσουν την αυσιπλοεία και την οικονομία κλπ. Άρα πρέπει να συμπαρασταθούμε στους Λιβύους, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, όλοι μας, τα κρατημέλη, οι θεσμοί μας, η χώρα που έχει την Προεδρία αυτή τη στιγμή, η Μάλτα, η χώρα μου δηλαδή, όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν για το σκοπό αυτόν. Έλεγα όμω για την Μεσόγειο εν γέννη. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μεσόγειο είναι άμεση και έμεση επίπτωση των όσων συμβαίνουν και στη Λιβύη αλλά και στην υπόχασα Αφρική. Πρέπει να βοηθήσουμε τις περιοχές αυτές να σταθούν στα πόδια τους οι άνθρωποι να αποκτήσουν δουλειές και έτσι να μην αντιμετωπίζουμε πλέον ούτε δύσκολους χειμώνες ούτε δύσκολα ε, καλοκαίρια στην, στην άμεση γειτονία μας. Πρόεδρος, σε η κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω γερμανικά για αλλαγή και πρέπει να σας πω ότι έχω μείνει λίγο άναυδη και λίγο συγκλονισμένη. Με βάση όλα αυτά που ακούμε, συζητούμε και με τον τρόπο που συζητούμε σήμερα. Θέλουμε να σώζουμε ζωές, δεν θέλουμε να πνίγονται οι άνθρωποι στη Μεσόγειο. Γι' αυτό δεν θα πρέπει κανένας να μπαίνει σε αυτά τα σκάφη, στις λιβικές ακτές. Αλλά αν δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, σε ποια στρατόπεδα, χωρίς τα ελάχιστα, ε, τα στοιχειώδη ε, από συνθήκες υγιεινής με διακίνηση, με καταναγκαστική εργασία, με αναγκαστική πορνεία, με βασανιστήρια, με ραπτισμούς, ξυλοδαρμούς, εκεί τους στέλνουμε ακούω ότι δεν θα πρέπει να ανεχθούμε να γίνει η Λιβύη μια αποτυχημένη χώρα. Fail state. Hello, είναι ήδη αποτυχημένη χώρα. Ε, κράτος διαλυμένο η Λιβύη. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να λειτουργεί. Ούτε σε ένα ελάχιστο της επικράτειας. Ακούω ότι υπάρχουν δύο εκτοφυλακές ε, που ε, αναφέρονται η μία στο ένα Υπουργείο και άλλη στο άλλο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει κανένας δημόσιος θεσμός, ούτε ακτοφυλακή, ούτε υπολείμματα οποιασδήποτε δημόσιας διοίκησης που να μην έχει διαποτιστεί από το οργανωμένο έγκλημα και τους εγκληματίες διακινητές. Και εμείς λέμε οι καημένοι Ευρωπαίοι που πληττόμαστε από τη μετανάστευση και την προσφυγιά να μείνουν εκεί, δεν τρέχει τίποτα. Αυτά που συζητούμε και ο τρόπος με τον οποίο είναι ανίποτα. Ωραία λόγια λέμε τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές για τις αξίες και τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προς Θεού να μην έρθει κανένας πρόσφυγας στην Ευρώπη. Και θα ε, εκπαιδεύσουμε, λέμε, μια ανύπαρκτη ακτοφυλακή και να τους κρατήσουν οπωσδήποτε στη Λιβύη, σε συνθήκες που ε, ακούμε και περιγράφουμε ε, όχι μόνο σήμερα. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Λιβύη Εντάξει, ευχαριστούμε την Υπηρεσία εξωτερική δράση για όσα κάνει, αλλά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Η διάλυση της Λιβύης άρχισε να μας ενδιαφέρει από τότε που είδαμε ότι υπάρχουν εκεί πολλοί πρόσφυγες που ενδεχομένω αύριο να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Προηγουμένως δεν ίδρωνε τα αυτή μας καθόλου για τη Λιβύη. Εδώ πολύ πολύ έτσι στο περιθώριο. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο και μια χρονική στιγμή που θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να συζητήσουμε πραγματικά τι κάναμε λάθος στο παρελθόν έτσι ώστε να βγάλουμε τα διδάγματά μας για το μέλλον. Διότι η Λιβύη δεν είναι η μοναδική αιστεία κρίσεων την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα να μην τη βοηθήσουμε καθόλου γιατί ακούω 90 εκατομμύρια ότι θα διαθέσουμε έτσι ώστε να υποστηριχθούν ε, δήμοι και κοινότητες και πολλά ακόμα. Και ποιες εγγύησεις έχουμε παρακαλώ ότι τα χρήματα θα πάνε ακριβώς εκεί που θέλουμε, όπου τα στέλνουμε. Ότι θα πάνε στο σωστό αποδέκτη και στο τελικό αποδέκτη που είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Ποιες εγγύησεις έχουμε ότι αυτά τα 90 εκατομμύρια που θέλουμε να βοηθήσουμε να στηθούν στα πόδια τους οι κοινότητες δεν θα ε, πέσουν σε χέρια εγκληματιών για να συνεχίσουν τις business με τους ε, πρόσφυγες όπως τις ξέρουμε. Και μήπως δεν πρέπει να αναζητήσουμε άλλη εναλλακτική πρόταση για τους πρόσφυγες χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση. Να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους στη Λιβύη να σταθούν στα πόδια τους. Εγώ πραγματικά έχω συγκλονιστεί από αυτά που ακούμε ότι δίνουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, με μια συμφωνία τύπου Τουρκίας με τη Λιβύη στο προσεχές μέλλον. Με όσες επικρίσεις και αν έχουμε προς την Τουρκία και μάλιστα και τα τελευταία αυτά γεγονότα, εν πάση περιπτώσει εκεί λειτουργεί η κυβέρνηση. Στη Λιβύη δεν λειτουργεί τίποτα. Και το θεωρώ πραγματικά ντροπή Έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια κατοίκους. Είμαστε πλούσια ήπειρος. Ε, έχουμε μια ευημερούσα Ευρώπη και κατά τα άλλα επιπολαιότητα. Λεφτά να σας δώσουμε, αλλά δεν έχουμε να σας προσφέρουμε τίποτα άλλο. Πραγματικά έχω μείνει άναυδη και έχω συγκλονιστεί ότι συζητάμε να αφήσουμε ε, στη Λιβύη τους πρόσφυγες αυτούς τα επόμενα δύο-τρία χρόνια με τη δικαιολογία ότι θα δώσουμε τίποτα κονδύλια. Εντάξει, δεν είναι λίγα τα 90 εκατομμύρια, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά από εκεί και πέρα ανεχόμαστε να ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε αφόρητες συνθήκες και μετά χαλαρώνουμε, ξεχνάμε τους πρόσφυγες γιατί δεν είναι στην Ευρώπη και μάλιστα δικαιολογούμε και τη συνείδησή μας ότι έχουμε κάνει κάτι. Όλα αυτά τα βρίσκω απολύτως απαράδεκτα και αφόρητα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you. Ε, Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Και τώρα η φιλελεύθερη Σοφή Ιντεβέλτ. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Γιατί δεν υπάρχει συντονιστή. Η κυρία Γκρισπέκ δεν είναι εδώ. Κυρία Ιντεβέλτ. Να μιλήσω, βεβαίω. Εκ μέρου τη ομάδα μου. Ε, αλλά σε προσωπική βάση, βεβαίω. Οι επικεφαλείς κυβερνήσεων που πιστεύουν ότι είναι καλό να έχεις ε, παρεδώσει με την Λιβύη, ε, ας πάνε να δουν τι γίνεται και μετά θα τους ρωτήσουμε ξανά αν ε, είναι τόσο καλή ιδέα όντως. Εμείς είχαμε μια συμφωνία με τη Λιβύη το 11, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπερλουσκόνη έδωσε 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Λιβύη για τον ίδιο σκοπό που συζητούμε σήμερα. Δεν μάθαμε το μαθημά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο τίτλος νομίζω ότι είναι εξαιρετικά παραπλανητικός. Μας λέει ανθρωπιστικές επιπτώσεις επίκως, της πολιτικής μας. Υπάρχουν πολλά στραβά βεβαίως, αλλά το αποτέλεσμα αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αποτέλεσμα των δικών μας πολιτικών, των δικών μας επιλογών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι εικόνες οι ιστορίες είναι ανατριχιαστικές. Πήραμε μια άλλη έκθεση σχετικά με τις συνθήκες των ετούντων άσυλων, των προσφύγων, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο Πάπας, τον οποίο δεν αναφέρομαι και πολύ συχνά, αλλά είπε για τα ελληνικά στρατέποδα, αναφερόμενος σε αυτά ως στρατόπεδα συγκεντρώσεως ε, και ξεσκώθηκε ολόκληρη συζήτηση για τον όρο που χρησιμοποίησε, αλλά οι συνθήκε αυτέ είναι. Όχι μόνο στη Λιβύη, στη δική μα Ήπειρο, στην Ευρώπη. Οι συνθήκε αυτέ είναι ανατριχιαστικέ, είναι απαράδεκτε. Χθε μόλι ε, διάβαζα μια άλλη ιστορία για γυναίκε, κορίτσια, κορίτσια τεσσάρων ετών που βιάζονται συστηματικά. Φαντάζεστε να ήταν η κόρη σα. Αυτά συμβαίνουν σήμερα, εξ ονόματό μα, στην Ευρώπη. Και ξέρω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον υπάρχει μια στοιχειώδη συνέντευξη σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η λύση και την υποστηρίζουν φαντάζομαι όλοι. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Το Συμβούλιο Επικεφαλής Κυβερνήσεων και Κρατών μιλούν γι' αυτό και υποτίθεται ότι ενεσδούν και προτείνουν λύσεις. Θα πρέπει να ντρέπονται. Θα πρέπει να ντρέπονται και ιδιαίτερα επικεφαλής των κυβερνήσεων. Λυπάμαι, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν εδώ, αλλά οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων μας μιλούν για τις χριστιανικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά όλα γίνονται στο όνομα των, τι, των ε, χριστιανικών αξιών, δεν νομίζω. Αυτό είναι το φρούριο Ευρώπη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής, του φρουρίου Ευρώπη. Μπορούμε να μιλάμε όσο θέλετε για την εκπαίδευση της εκτοφυλακής του λιμενικού κλπ. Να τους λέμε για τη σύμβαση της Γενέβης Μα κοροϊδευόμαστε. Είναι επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι ή τι είναι η σύμβαση της Γενέβης. Όλα τα ξέρουμε, απλώς δεν μας νοιάζει. Και στο τέλος τι κάνουμε, κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτήν την κατάσταση. Και δεν είναι δυνατόν η πολιτική για το άσυλο να γίνει κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, γιατί τότε έχει ξεφύγει από τα χέρια μας. Ο κ. Ποντιρόλη είναι εδώ, αλλά δεν είναι δικό σας το θέμα, κ. Ποντιρόλη. Το θέμα είναι ότι διολυσθένει η πολιτική για το άσυλο σε μια, προς μια περιοχή για την οποία δεν έχουμε κανέναν λόγο. Ε, και μάλιστα λόγω δεν έχουν ούτε καν τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει να αντισταθούμε λοιπόν, να δώσουμε μάχη σκληρή σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι πολιτικές αυτές να παραμείνουν ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να θεραπεύσουμε αυτήν την κατάσταση, να δώσουμε τέλο ε, στα βάσανα αυτών των ανθρώπων. Να δώσουμε μια αξιοπρεπή λύση στο πλαίσιο μια ενιαίας πολιτική μετανάστευση και για το άσυλο. Και το λέω αυτό από την αρχή. Οι επικεφαλής των κυβερνήσεων, οι αρχηγοί κυβερνήσεων που πιστεύουν ότι αυτό είναι λύση, να πάνε να μείνουν λίγο σε αυτά τα στρατόπεδα και μετά να μας πούν πραγματικά τι πιστεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Η κυρία Γιούντιτ ε, Σαρχεντίνη, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Οι εκπρόσωποι των γιατρών μάλλον η εκπρόσωπος των γιατρών χωρίς σύνορα ρώτησε κάτι ε, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και χρειάζεται απάντηση ότι η λύση δεν είναι να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτό το σύστημα. Το αντίθετο, θα χρηματοδοτηθούν ακόμα περισσότερο οι στρεβλές αυτές ε, καταστάσεις. Δεν άκουσα απάντηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων μας και πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται, γιατί εκεί είναι η μεγάλη διάσταση των απόψεων. Ε, εκτός του γεγονότος ότι η καταπολέμηση της διακίνησης ε, προσπαθώντας να συλλάβουμε ε, τους διακινητές δεν σημαίνει ότι θα εκριζωθεί και θα εξαφανιστεί η διακίνηση. Ε, κάνουμε εδώ μια περίεργη συζήτηση στην Επιτροπή Ελευθεριών. Ακούμε ε, διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές πραγματικότητες και προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Ούτε πρόκειται να ε, πετύχει η πολιτική μας αν εφαρμόσουμε αυτά που νομίζουμε ότι είναι πραγματικότητα. Λέτε ότι ε, εκπαιδεύουμε την ακτοφυλακή της Λιβύης, το λιμενικό τους και τους μαθαίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη, μάλιστα. Τα κέντρα κράτησης δεν υπάγονται στην ακτοφυλακή, δεν υπάγονται σε κανέναν βασικά, το καν στο κράτος. Και όταν μας μιλάτε για τις λιβικές αρχές στον πληθυντικό, αυτό είναι αστείωτητα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Δεν υπάρχουν οι αρχές. Το πληθυντικό μάλιστα είναι οι αρχές. Δεν ξέρουμε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Και ποιος παίρνει αποφάσεις για τα κέντρα κράτησης, πώς υλοποιούνται. Και στα χέρια ποιας αρχής είναι αυτά ή ποιον αρχών στο πληθυντικό. Είναι τελείως άναρχα. Χάνουμε πραγματικά ε, το στόχο μας εδώ. Άκουσα την Birgit να μιλούν και τη Σοφία Νιτβέλτ. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπαν, αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε και να καταλάβουμε τι είναι αποτελεσματικό και τι δεν είναι. Και μέχρι στιγμής το να αφήνουμε τους Λιβύους να διασώζουν εντό εισαγωγικό κόσμο από τη θάλασσα και να τους πηγαίνουν στη στεριά, δεν σημαίνει ότι τους σώζουν. Σημαίνει ότι επιστρέφουν οι άνθρωποι αυτοί σε άλλα κολαστήρια που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αυτά. Και το πρώτο που είπε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν εάν αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται πρόσφυγε ή μετανάστες. Αυτό μας μάρανε. Αυτό είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βοηθούμε ε, με την τακτική μας ή υποδαβλίζουμε ε, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ τελευταίο συντονιστή. Είναι συντονίστρια κυρία Φεράρα από την ομάδα EFTD. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί στις 4 κανονικά αρχίζει το επόμενο θέμα μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να επιζητούμε μία συνεργασία και εταιρική σχέση με τη Λιβύη είναι κάτι το σουρεαλιστικό. Ε, μιλήσαμε και για τη συμφωνία με την ε, Τουρκία, την οποία καταγγείλαμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι το αποδοτικό ως προς τα αποτελέσματα. Και είναι και επιβλαβές ως προς τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τις διαδικασίες και την τήρηση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως προς την τελική επαλήθευση της χρήσης αυτών των χρημάτων. Γιατί και οι γιατροί χωρίς σύνορα μας επιβεβαιώνουν ότι δεν θα λυθούν τα ζητήματα χορηγώντας ακόμα δεν τα ζητήματα χορηγώντας περισσότερα χρήματα. Είναι ένα ενδυμικό θέμα το οποίο δεν θα επιληθεί με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε μετά τη συμφωνία με την Τουρκία ότι οι αποβιβάσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί, αλλά έχουν αυξηθεί στην Ιταλία. Και αυξήθηκαν και οι θάνατοι κατά συνέπεια. Άρα θα πρέπει να προβάλλουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Θα ήθελα μία απάντηση λοιπόν στο ερώτημά μου είτε από την ΕΕΔ είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται μία συζήτηση τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις υπηρεσίες διάσωσης και έγινε και μία ακροαματική διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα και των εισαγγελικών αρχών της Κατάνια σε σχέση με το ρόλο και της Frontex και των ΜΚΟ. Δεν θέλουμε να γενικεύουμε, θέλουμε να γίνεται όμως διάκριση μεταξύ ΜΚΟ που εργάζονται υπό συνθήκες διαφάνειας και μήκυο που δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε από πού χρηματοδοτούνται, όπως είπε και ο εισαγγελέας της Κατάνια. Και φαίνεται ότι ε, υπάρχουν επαφές με λιβικές αρχές φέρουν, δηλαδή φορούν τις στολές της ε, ακτοφυλακής, αλλά δεν είναι άνθρωποι της ακτοφυλακής της Frontex. Και αυτό αφορά τη δράση στα δυτικά παράκτια της Λιβύης. Γίναμε, έγινε λόγος για τον Τρίτονα, τη Σοφία, το, τη U4Med και συμφωνίες με χώρες που δεν είναι καθόλου σταθερές. Τι έλεγχος υπάρχει επί της ουσίας σε σχέση με τα λεγόμενα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Frontex. Ποιες είναι οι σχέσεις ΜΚΟ, συγκεκριμένων ΜΚΟ, με την δίθεν ακτοφυλακή της Λιβύης. Ωραία. Τέσσερις. Τέσσερις ακόμα θα λάβουν το λόγο. Θα ήθελα να περιοριστείτε στα ένα-δύο λεπτά. Κυρία Κίνγκε. Ευχαριστώ. Με λυπεί να βλέπω αυτές τις εικόνες, πραγματικά. Είναι κάτι το τρομακτικό. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι προσπαθούμε ε, και πολλές φορές συλλαμβάνουμε ανθρώπους και αυτό εξαρτάται από το, από το χρώμα του δέρματός τους. Δηλαδή, ε, πολλές φορές συλλαμβάνονται άνθρωποι επειδή δεν είναι λευκοί. Αυτό το έκανε και ο Καντάφη και το συνεχίζουν και σήμερα οι Λιβικές αρχές επίσης το εμπόριο οργάνων υπάρχει στη Λιβύη, εκτός και εντός κέντρων. Και αυτά δεν τα βλέπουμε εδώ. Η Επιτροπή και η ΕΡΙΕΔ είπε ότι δεν εργαζόμαστε μόνο για τους μετανάστες, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που έχει καταρακωθεί κοινωνικά. Πρόκειται για ένα μη κράτος Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν για αυτούς που παραμένουν σε αυτά τα κέντρα, ποιος ε, θα επιβιώσει και ποιος θα φύγει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να επανεγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς το αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί είναι απαράδεκτο να μην σώζονται ζωές τη στιγμή που η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό. Πώς χειριζόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μιλάμε λοιπόν να, το να βρεθούν οι άνθρωποι σε αυτά τα κέντρα, αλλά να διαφύγουν από τη Λιβύη. Η Λάουρα Μίλησε και για την κατάρτιση της ακτοφυλακής. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση και επαναλαμβάνω και εγώ την ερώτηση. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτά που προανέφεραν οι συνάδελφοι. Στη ε, Λιβύη η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την Τουρκία. Άρα δεν μπορούμε να προτείνουμε τα ίδια μέτρα. Αλλά αυτός θα πρέπει να είναι ο απότερος στόχος μέσα στα πλαίσια ε, μίας ε, γενικότερης συμφωνίας. Γιατί όπως είπε η Λάουρα Φεράρα, με τη συμφωνία με την Τουρκία στην ουσία κλείσαμε την οδό των ε, Βαλκανίων και έχουν, έχουν αυξηθεί οι αποβάσεις στις Ιταλικές αρχές. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και ορισμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν σε σκέψη. Τη στιγμή δηλαδή που η Ραγούζα και οι Σιρακούσες μας έδωσαν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για το Ποτσάλο και την Αουγκούστα, αυτές, αυτούς τους δύο λιμένες όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Μόνο το 5% εκείνων που φτάνουν στη Σικελία αφορούν τις νέες ε, ε, εθνοτικές μειονότητες οι οποίες εντάσσονται στο σχέδιο επανεγκατάστασης, δηλαδή σε σχέση με ένα 5% και αυτό αφορά το, τα στοιχεία του 17 σε σχέση με το 16. Αυτό που έχει σημασία είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορούμε να δεχτούμε στη Λιβύη να υπάρχουν αυτές οι αποτρόπες συνθήκες οι οποίες ε, προαναφέρθηκαν παράλληλα, όμως θα πρέπει να προβάλλουμε μία βελτίωση των συνθήκων ζωής ε, στις αφρικανικές χώρες, όπου επικρατούν άθλιες οικονομικές συνθήκες, αλλά επαναλαμβάνω ότι εδώ ε, δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις σε σχέση με περιοχές που ζουν μία εμπόλεμη κατάσταση και από εκείνες τις περιοχές προέρχονται οι πρόσφυγες. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε όλες τις μεταναστευτικές ροές, αδιακρίτως. Ο κύριος Δεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά θα είμαι σύντομος γιατί είπαν πολλά οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα των σοσιαλιστών δημοκρατών, των πρασίνων και των φιλελευθέρων και με κάλυψαν. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες εβδομάδες είδα ένα διαπιστευμένο έγγραφο που περιέγραφε την κατάσταση στη Λιβύη ως ε, τελείως απελπισμένη και απελπιστική. Ε, ότι δεν μπορεί κανείς να προσπαθήσει να κάνει τίποτα, ούτε για τα κέντρα κράτησης, ούτε για την προστασία των ακτών, ούτε τίποτα. Ένα το συμπέρασμα ότι είμαστε τελείω ανήμποροι. Μίλησα και με εκπροσώπου του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση πριν από λίγε εβδομάδε και μα είπαν ότι στο προσεχέ μέλλον μάλλον δεν θα γίνει τίποτα. Και επίση, γιατί μεταξύ άλλων, ένα λιβικό δικαστήριο ε, ακύρωσε ή επεφάθη ότι ήταν άκυρη η συμφωνία Λιβύης-Ιταλίας. Ακόμα και αν θέλαμε να κάνουμε μια συμφωνία με ένα αποτυχημένο κράτος, οι δικοί σας εμπειρογνώμονες λέγεται ότι δεν γίνεται. Γιατί να συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο που προκαλεί μόνο δεινά. δεύτερο. Όταν ακούμε ότι είναι η κατάσταση πολύ ε, άσχημη και φρικτή στην ε, Λιβύη, γιατί δεν το πάμε δίπλα στην Ισία ή στο Μαρόκο, αφού με το Μαρόκο έχει ήδη συμφωνία η Ισπανία. Να μεταφέρουμε δηλαδή το πρόβλημα από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτό το θεωρώ απολύτως επικίνδυνο. Όταν αρχίζουμε να διαρευνούμε και τέτοια ενδεχόμενα που δεν είναι λύσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, την Ισία. Και τέλος, από όλη αυτή την ιστορία, Εμένα μου λείπει αναφορά στην πολιτική της είπα της αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Δηλαδή, από ανθρωπιστικής ε, απόψεως, η μόνη λύση θα ήταν να δοθεί πρωταγωνιστικός ρόλος στην ύπατη αρμοστία, ιδιαίτερα για τη μετεγκατάσταση. Γιατί από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Υπάρχουν προγράμματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα λοιπά που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τουλάχιστον κάπως να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ε, ε, ο κύριος Βάιντεν Χολτσερ, έχω μια σύντομη ερώτηση προς το πάνελ. Πώς φαντάζεστε την κατάσταση σε ένα, δύο, τρία χρόνια από σήμερα, αν συνεχιστεί δηλαδή ε, αυτό που επικρατεί εκεί, τι προβλέπετε να γίνει. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην το ανεχθούμε αυτό εδώ στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο, να δραστηριοποιηθούμε πολύ περισσότερο, να φωνάξουμε πολύ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι απολύτως απαράδεκτα που ακούμε. Και έχουμε υποχρέωση ως εκλεγμένοι προσωποί των ευρωπαϊκών λαών να ε, είμαστε ε, ενεργοί βουλευτές δραστήριοι, να φωνάξουμε, αλλιώς θα έχουμε και εμείς ευθύνη και θα είμαστε και εμείς ένοχοι. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε και πολλέ ερωτήσει. Ο κ. Παντηρόλη από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Καθώ ο χρόνο πιέζει πολύ γρήγορα, θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποιε από τι ερωτήσει και να σχολιάσω κάποια από τα σχόλια. Πολλοί αναφερθήκατε στο θέμα των συνθήκων στα κέντρα κράτησης και το τι να έχει να σώζουμε ζωές για να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα στρατόπεδα. Κοιτάξτε, σώσαμε 35.000 ανθρώπους. Ε, αυτοί που διασώζονται σε ευρωπαϊκά ύδατα πηγαίνουν στην Ιταλία. Δεύτερον, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είναι νέα ιστορία. Η Λιβική εκτοφυλακή πέρσι μέσωσε χιλιάδες ανθρώπους όμως ξέρετε ότι υπάρχουν από 700.000 έως 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Λιβύη, ε, πολλοί σε αυτά τα στρατόπεδα και όπως είπατε και πολλοί από εσά. Ε, υπάρχει πολύ χρήμα πίσω από αυτήν την ε, υπόθεση. Υπάρχουν οι δουλέμποροι. Λοιπόν, χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μιλάμε για αυτό που κάνουμε στον Ήγηρα, στο Τσάντ, στην Νότιο Λιβύη, για να σταματήσουμε ακριβώς την παρανομή μετανάστευση, ε, δεν εφαρμόζουμε μόνο ελέγχους στα σύνορα. Έχουμε και προσφέρουμε και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις, γιατί πολλές από τις κοινότητες αυτές που ζουν στον δρόμο της μετανάστευσης, οικονομικά ζουν και κερδίζουν, θα μάλιστα, από την διακίνηση αυτή των μεταναστών. Άρα δεν πρόκειται, και σίγουρα δεν είναι αυτό η πρόθεσή μα να ενισχύσουμε του ελέγχου στα σύνορα. Δεν γίνεται έτσι. Γίνονται πολλέ προσπάθειε στην Νότιο Λιβύη, που δεν είναι και εύκολα προσβάσιμη να ξέρετε, και στι χώρε νοτίω τη Λιβύης και για του ελέγχου στα σύνορα, αλλά και, και κυρίω θα έλεγα, στον οικονομικό τομέα προσπαθούμε να προσφέρουμε εναλλακτικέ απασχολήσει σε αυτού του νέου ανθρώπου που δουλεύουν στο δουλεμπόριο, στο οποίο, όπω είπα, υπάρχει πολύ χρήμα. Τώρα, όσον αφορά τα κέντρα, τα κέντρα κράτηση, όπω είπε και ο κύριο Παπόφσκι, η άμεση προτεραιότητά μα είναι να βελτιώσουμε τι συνθήκε. Σήμερα, τώρα. Μακροπρόθεσμα όμω, ο σκοπό είναι να δημιουργήσουμε εναλλακτικές εγκαταστάσεις που δεν θα είναι υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων. Έξω λοιπόν σημαντικό είναι ενίσχυση, η ενίσχυση της παρουσίας μας στην Λιβύη. Ήμουν και πήγαν και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι στην ε, Λιβύη. Μίλησαμε με τις τοπικές αρχές, μίλησαμε με τους ανθρώπους. Αλλά και πάλι όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι θα λύσουμε το πρόβλημα αύριο. Υπάρχουν πολλά άλλα, πολύ περισσότερα που πρέπει να κάνουμε. Οπότε η μακροπρόθεσμη λύση είναι οι άνθρωποι να φύγουν από αυτά τα κέντρα. Είτε να παραπατριστούν με κάποιο σύστημα επιστροφής, είτε να εξεύρουμε μακροπρόθεσμες λύσεις για την κράτηση, την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων στη Λιβύη. Όσον αφορά την κατάσταση, δύο-τρία χρόνια από σήμερα, δεν έχω γυάλινη σφαίρα, αλλά τι να σας πω, η γενικότερη οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται και μάλιστα ταχύτατα και μάλιστα θα έλεγα που οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα προς την καταστροφή. Διότι η Λιβύη εξαρτάται σχεδόν 100% από τις εξαγωγές πετρελαίου, οι οποίες έχουν καταρρεύσει, έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου και δεν φαίνεται να ευρίσκονται εναλλακτικές λύσεις τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Είναι κακή λοιπόν η οικονομική κατάσταση, έχουμε στασιμότητα και ύφεση. Τα μέρη πρέπει να ξέρουν μια από κοινού λύση. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τα κράτη-μέλη, δουλεύουμε με τον Αφρικανικό Σύνδεσμο, με την Ένωση Αφρικανικών Κρατών, με την Αίγυπτο κλπ. Και όσον αφορά την ασφάλεια τώρα, και εκεί η κατάσταση επιδεινώνεται. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει αμέσως και εμέσως τις αντιμεχόμενες παρατάξεις. Έχουμε εγκληματικότητα, απαγωγές. Γι' αυτό και οι προσπάθειες δεν αποδίδουν άμεσα. Χρειάζεται λοιπόν φυσική ε, παρουσία. Εμείς είμαστε εκεί. Τα Ηνωμένα Έθνη για να καταλάβετε δεν είναι στη Λιβύη θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί εν μία νυχτή και σίγουρα όχι αύριο. Μια ερώτηση που δεν νομίζω ότι απαντήθηκε, λέει κύριε Σαρζεντίνη, και νομίζω ότι την ακούσατε, αλλά την παραλείψατε. Να την παραλάβω. Θέλω μια απάντηση, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης. Γιατί η κυρία από του είπε η χρήση πόρων από το φρύγιο Ταμείο ουσιαστικά τι κάνει, ρίχνει περισσότερα χρήματα σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ενισχύει ακριβώς τους δουλεμπόρους. Ουσιαστικά ενθαρρύνουμε έτσι εν τέλει τα ανθρωπιστικά προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Και Ποπόφσκι. Ο κ. Ποπόφσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δυστυχώ έχει πέρασει η ώρα αλλά η χρηματοδότηση που προσφέρουμε εμεί δεν απευθύνεται ούτε στην κεντρική τράπεζα ούτε στην κεντρική κυβέρνηση τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει τη διεθνή εταίρους. Πρώτη είναι είπα αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγες και τη χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα χωρίς αυτή. Ή ο διεθνή οργανισμό μετανάστευση. Θα πρέπει να επανέλθουν οι ε, οργανώσει εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό δεν εξαρτάται από εμά. Εμεί συνεργαζόμαστε από εταίρου αξιόπιστου, που έχουν αποδείξει στην πράξη την ε, αξιοπιστία τους. Ο συνομιλητή και ο αποδέκτη των χρημάτων λοιπόν δεν είναι η Λιβική κυβέρνηση, ούτε προτιθέμεθα να κάνουμε καμία συμφωνία με τη Λιβική κυβέρνηση. Και κατά τα άλλα, εμεί συνεργαζόμαστε μόνο με την κυβέρνηση τη Εθνική Ενότητα που αναγνωρίζεται για κάποια αντίστοιχη συμφωνία με την ε, Τουρκία. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στις λιβικές αρχές στον πληθυντικό, αυτό αφορά τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι κάποιες ε, αρχές που λειτουργούν και κάποιες στοιχειώδεις υπηρεσίες τις παρέχουν. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. και τα όσα μας περιγράψατε. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί στις 3 Μαΐου με ε, παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, των αντίστοιχων θεμάτων και ε, επίσης θα ακούσουμε και την έκθεση της Επιτροπής που πήγε την περασμένη εβδομάδα στην Ιταλία. Και θα τη συνδυάσουμε με ανταλλαγή απόψεων με τον Ιταλό Υπουργό Ιστορικών. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι. And, uh... Ευχαριστώ να πάτε στο καλό μου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Online, ε, we start ε, the point. Στις 9 Μαρτίου του 2017, και στο σημείο 5, η Ευρωπόλ δημοσίευσε την έκθεσή της για το 2017 σχετικά με την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα. ΣΟΚΤΑ ονομάζεται η έκθεση αυτή. Στην εποχή της τεχνολογίας από το 2018 μέχρι το 2021 έχουμε ένα νέο κύκλο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Με στρατηγικούς στόχους που θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές δράσεις απέναντι στο σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα. Το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στην επόμενη συνεδρίασή του θα αποφασίσει ε, περί των νέων ε, προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση του έγκληματος για το επόμενο διάστημα. Σήμερα η Ευρωπόλ και ο διευθυντής της, ο κ. Ροπ Γουένραιτ, έχει έρθει να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Ε, οπότε είναι σημαντική ευκαιρία για μας να ανταλλάξουμε απόψεις. Παρακαλώ κύριε Γουένραιτ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω ότι έχουμε την λανθασμένη παρουσίαση. Θα ήθελα να γίνει διόρθωση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σήμερα να σας παρουσιάσω την πολιτική μας σε σχέση με την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι μια εμβληματική προσπάθεια και πολιτική και αποτελεί ακρογωνία λίθο για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ο κύκλος αυτός της πολιτικής καλύπτει την περίοδο από το 2018 μέχρι το 2021 και η έκθεση είναι η έκβαση της πιο συνεκτικής συλλογής αποτελεσμάτων για το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή 2.300 ε, ερωτηματολόγια από πολλές ε, οργανώσεις σε σχέση με τη συμμετοχή της Eurojust, ε, Europol, Interpol και Frontex είναι η πιο εμπεριστατωμένη έρευνα που έχει γίνει μέχρι τούδε σε σχέση με την προγενέστερη. Έχουμε το διπλάσιο αριθμό δεδομένων. Ένα βασικό στοιχείο των πολιτικών συζητήσεων στο Συμβούλιο θα βασιστεί σε αυτή την ε, αξιολόγηση για να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για την ε, επόμενη τετραετία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και φυσικά θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ιδιαίτερα οι οργανισμοί επιβολή των μέτρων μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων και επιχειρησιακών δράσεων για να μπορέσουμε να ε, αναχαιτήσουμε την, το οργανωμένο έγκλημα. Διαφάνειες παρακαλώ, λέει ο μιλητής. Ωραία, θα συνεχίσω χωρίς διαφάνειες. Σε σχέση με τις εγκληματικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 3.600 οργανωμένες ομάδες και τώρα φτάσαμε σε 5.000 φέτος. Και αυτό αντικατοπτρίζει τη σωστή δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και φυσικά ε, βλέπουμε ότι ανακύπτουν και μικρότερες ομάδες οι οποίες είναι αλληλένδετες και έχουν ε, νέα δυναμική, είναι, διαφοροποιούνται περισσότερο και μπορούν να προσαρμοστούν και να δράσουν σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Είχαμε 180 εθνικότητες και αυτό δείχνει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, τα έχουμε ε, ομάδες που απαρτίζονται από πάνω από μία εθνικότητα και βλέπουμε λοιπόν πώς ορίζονται από τη Europol. Επόμενη διαφάνεια ως προς τις ε, μεγαλύτερες απειλές, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι και το πιο σημαντικό, έχει αυξηθεί εκθετικά όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια και αφορά και το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν επιγραμμικά σε διάφορες επιχειρήσεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν εγκλήματα τα οποία συνδέονται με τον κυβέρνο χώρο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια υπηρεσία εγκλήματος, δηλαδή το έγκλημα ως υπηρεσία, το οποίο προσδίδει και τα κατάλληλα μέσα για να μπορεί να δημιουργηθεί μία αγορά εγκλήματος και φυσικά και εγκληματικές ικανότητες που γνωρίζουν όλο ένα και μεγαλύτερη εμβέλεια μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την τεχνολογία. Αυτό αφορά και ένα συγκεκριμένο λογισμικό, κρυπτολογισμικό που χρησιμοποιείται. Αφορά βεβαίως και την ε, χρησιμοποίηση των παιδιών και την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών ένα φαινόμενο που γνώρισε όλο ένα και αυξανόμενη εμβέλεια. Και πιστεύω ότι και αύριο θα σας μιλήσουμε για τη δραστηριότητα της Europol μέσα στα πλαίσια της ε, ακρόασής σας. Επίσης υπάρχει η υπηρεσία πληρωμών και εδώ ε, δρά το οργανωμένο έγκλημα. Βλέπουμε λοιπόν πώς, έχει το, πώς έχουν οι επιδραμικές δραστηριότητες σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών. Πώς δηλαδή χρησιμοποιούνται τα χρήματα, τα κονδύλια και πώς έχει η κατανομή, οι πλατφόρμες μάλλον κατανομής, ιδιαίτερα στο ε, Darknet, όπου χρησιμοποιείται για να πολιθούν φαρμακευτικά σκευάσματα και παραχαραγμένα προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υφίσταται αυτή η αγορά παράνομων αγαθών και υπηρεσιών και το 1% των χρηστών του Darknet είναι υπεύθυνο για το 50% των ε, χρηματικών συναλλαγών. Όμως ε, η μεγαλύτερη δραστηριότητα αφορά τα ναρκωτικά. Το 1 τρίτο της δραστηριότητας ε, αφορά ένα 75% ε, το οποίο σχετίζεται με την εμπορία ενός ή περισσότερων ειδών ναρκωτικών και φυσικά το Darknet είναι εκείνο το οποίο προωθεί όλα τα είδη ναρκωτικών. Βλέπουμε λοιπόν μία αύξηση της ε, χρήσης της κανάβεως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα περισσότερα είδη κανάβεως προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Και ιδιαίτερα στη Λιβύη υπάρχει μεγάλη καλλιέργεια μέσα στα πλαίσια της αφρικής και η κοκαίνη χρησιμοποιείται και εμπορεύεται, αλλά ιδιαίτερα ως προς τα σύνθετα ναρκωτικά βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε συνθετικά ναρκωτικά βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με νέες τεχνικές παραγωγής και νέες ουσίες πάνω από 400 ουσίες οι οποίες έχουν ανεχνευθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επίσης, έχει αυξηθεί και η ικανότητα παραγωγής των συνθετικών ναρκωτικών και φυσικά μια μεγάλη παραγωγή και ένα πολύ ευρύ δίκτυο διανομής. Εδώ μιλάμε για το έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, διαρρήξης σε σπίτια, οχήματα και εδώ βλέπουμε ότι οι ομάδες αυτές δρούν ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και πολλές φορές μιλάμε για μικροέγκλημα, μικροεγκλήματα, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα έγκλημα ευρείας εμβέλειας, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για οργανωμένο έγκλημα. Οι διαρρήξεις έχουν αυξηθεί άρδιν τα τελευταία χρόνια και αφορά όχι μόνο τις οικίες αλλά και τις επιχειρήσεις οι διαρρήκτες χρησιμοποιούν επιγραμμικά, επιγραμμικά συστήματα και στα δίκτυα κοινωνικής ε, δικτύωσης προσπαθούν να φτάσουν σε μία στοχοθέτηση συγκεκριμένων ε, περιοχών σε σχέση με τα μέσα που διαθέτουν για την εγκληματική αυτή δραστηριότητα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι μας ενδιαφέρει και το ε, περιβαλλοντικό έγκλημα, δηλαδή η διακίνηση αποβλήτων και απορριμμάτων καθώς και ε, ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η διακίνηση φυσικά των μεταναστών είναι μία ολοένα διονγκούμενη αγορά και αφορά μια μεγάλη κατηγορία με πολλές ομάδες διακινητών. Μιλάμε για 3 με 5 δις έσοδα. Και φυσικά ε, χρησιμοποιείται και, το, και μια πλατφόρμα όπου συμμετέχουν πολλοί υποφορείς σε σχέση και με το ξέπλυμα Ευρώμικου χρήματος, ε, της ε, διακίνησης, της εκμετάλλευσης παιδιών και ούτω καθεξής. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της διακίνησης ε, μεταναστών με την παράδοση παράνομων εγγράφων και παραχαραγμένων εγγράφων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ε, ροή, υπήρχε μία ροή από την Ανατολική στη Δυτική Ευρώπη, αλλά τώρα υπάρχει μία νέα δυναμική προς όλες τις κατευθύνσεις και αφορά και την εκμετάλλευση στον τομέα της εργασίας. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την, ε, δυστυχώς το, τα συνόδευτα παιδιά, τα οποία ε, μπορούν ε, δυστυχώς να χρησιμοποιηθούν για την εμπορία οργάνων. Επίσης, οι διακινητές χρησιμοποιούν τη τεχνολογία και τα, την κοινωνική δικτύωση σε όλα τα στάδια της εγκληματικής δραστηριότητας. Δηλαδή, η τεχνολογία συνδράμει σε όλους αυτούς τους τομείς. και όπως γνωρίζετε οι, τα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν ολοένα και μία διονγκούμενη αγορά έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν αυτά τα χρήματα στην νόμιμη οικονομία. Αυτό το ξέπλυμα αφορά και μία ειδική τεχνογνωσία και τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα στα πλαίσια ε, τάχιστων συναλλαγών και διαδικασιών τάχιστης νομιμοποίησης έτσι ώστε ε, αυτά τα έσοδα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα. Πολλές φορές εμβάζονται χρήματα και δεν υπάρχει σωστός έλεγχος από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Γι' αυτό θα πρέπει οι αρχές να ε, πατάξουν αυτό το έγκλημα. Ε, ξέρετε ότι το, τα μετρητά δεν χρησιμοποιούνται πλέον τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά και τα μετρητά ακόμα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής εγκληματικής δραστηριότητας. Μέσα στα πλαίσια του ξεπλήματος αυτού υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι, πολλοί μεσάζοντες και ε, συστήματα μεταφοράς χρημάτων τα οποία ε, δεν μπορούν να ανοιχνευτούν ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με prepaid cards. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολυσχηδές ε, μέσον χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνεται και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τέλος, Αυτό που έχουμε περιγράψει είναι ένας αριθμός απειλών και όλες αυτές οι απειλές είναι σημαντικές, αλλά ο, ρόλος της Europol είναι να μπορέσει να ορίσει τις πιο επικίνδυνες μορφές οργανωμένου εγκλήματος με βάση τα κριτήρια διαφάνειας μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΣΟΚΤΑ. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία έχουμε οκτώ προτεραιότητες για να αντιμετωπίσουμε τις πιο απειλητικές μορφές σοβαρού και επικίνδυνου εγκλήματος. Μιλάμε για το ε, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τα ναρκωτικά, την ε, διακίνηση μεταναστών, το οργανωμένο έγκλημα στις ιδιοκτησίες και φυσικά την διακίνηση ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει μία συνδεσιμότητα του οργανωμένου εγκλήματος, μία διασύνδεση όλων των τομέων. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοδότηση του εγκλήματος και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την παραχάραξη τεκμηρίωσης, καθώς και την ε, επιγραμμική, το επιγραμμικό εμπόριο παράνομων αγαθών και υπηρεσιών. Η τελευταία διαφάνεια δείχνει ποιες είναι οι βασικές απειλές και αυτό για να σας καταδείξουμε ποιοι είναι αυτοί οι τομείς συνολικά και υπάρχουν και ορισμένες υποκατηγορίες που είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όπου υπάρχει όλο ένα και διονγκούμενη δραστηριότητα. Επίσης, η παραχάραξη εγγράφων ε, προσλαμβάνει πολύ σημαντικό χαρακτήρα με βάση την διακίνηση των μεταναστών και των προσφύγων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να προσπαθήσουμε με βάση την εφαρμογή του νόμου να δούμε ποιες είναι οι πιο ε, απειλητικές μορφές οργανωμένου εγκλήματος έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις για να δράσουμε από κοινού έτσι ώστε με τα περιορισμένα μας μέσα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι συντονιστές παρακαλώ. Έχετε ερωτήσεις, ε, σχόλια. Ε, δύο λεπτά για τον καθένα. Μετσόλα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Wainwright, ο οποίος ε, περιδιάγραψε αυτά τα οποία έχει εντοπίσει η Europol στο πλαίσιο της τελευταίας μελέτης. Το ΕΛΚΑ ε, σας ευχαριστεί για την εξαιρετική σας δουλειά, για το ότι μας κρατάτε όλους ασφαλείς. Θα ήθελα να καλέσω τα κράτη-μέλη τώρα να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τακτικές στα συμπεράσματα της ε, μελέτης για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Ε, θα ήθελα να χαιρετήσω επίσης τις προτεραιότητες ε, για την περίοδο 18-21 που καταγράφονται στην έκθεση ΣΟΚΤΑ. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα προτιμούσα να είχα δει μεγαλύτερη έμφαση στην, στον αγώνα κατά της διαφθοράς στα κρατημέλη. Να προσθέσω ότι χθε στη χώρα μου, στην Μάλτα, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους ε, δρόμους λόγω φημών ότι ο Πρωθυπουργό και η οικογένειά του ήλεγχαν μυστικές εταιρείε στον Παναμά για διάφορες ε, παρανομές με το Αζερβαϊτζάν. Η θεσμική κρίση που αντιμετωπίζει η Μάλτα σήμερα είναι χωρί προηγούμενο. Και μάλιστα επιδρώνεται από το γεγονό ότι η αστυνομία στην Μάλτα ενήργησε με βάση οδηγίε από τον Πρωθυπουργό και έτσι πολύτιμο χρόνο, πολύτιμε ώρε χάθηκαν από τη στιγμή που μαθεύτηκαν τα γεγονότα ω την επέμβαση τη αστυνομία. Αυτά τα οποία έγιναν ήταν ε, πίστευτα ο κόσμος ε, τρέχει στις ε, τράπεζες πριν η αστυνομία επέμβει για να διασώσει τα στοιχεία. Η Europol λοιπόν επαναλαμβάνω κατακλείδη ότι πρέπει να κάνει προτεραιότητα τη διαφθορά. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω του πολίτες μας ότι είναι προτεραιότητα για σας τη διαφθορά και η ερώτησή μου είναι τι χρειάζεται η Europol για να μπορέσει να λάβει αγώνα διασυνοριακό κατά τη διαφορά χωρί την συνεργασία τη συνένεση αναγκαστικά των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικές ερωτήσεις. Αν δούμε το κατάλογο που μας παραθέσετε, ε, το είδος του εγκλήματος περί το οποίο συζητούμε δεν είναι τίποτα καινούριο, αλλά Κάθε φορά βλέπουμε ότι οι εγκληματίες βρίσκουν τον τρόπο να οργανώνονται ε, σε νέους τομείς, μετά επανέρχονται στους παλιούς, αλλά παραμένουν τα προβλήματα με το κοινό έγκλημα εντό εισαγωγικών, περισσότερα από τα προβλήματα που έχουμε με κάθε είδους τρομοκρατία. Είπατε ότι η συλλογή στοιχείων και η ανάλυση τους ήταν μεγαλύτερη ε, σε όγκο αυτή τη φορά όπως το παρελθόν και θέλω να ρωτήσω, συμμετείχαν πραγματικά όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχουν διαφορές. Βεβαίω είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές γιατί οι προκλήσεις αυτές δεν είναι ίδιες σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά με ποιον συνεργαζόμαστε, με ποιον είμαστε σε επαφή όταν προσπαθούμε να πετάξουμε αυτό το έγκλημα. Και επίσης, έχετε διαπιστώσει αλλαγές στην οργάνωση της δικαιοσύνη και της αστυνομίας ε, και στην τεχνολογία μαζί με τις νέες προτεραιότητες. Γιατί ακούμε και ιδέες για την αλλαγή στον τρόπο ε, δίωξης, έρευνας, συνεργασίας των δικτικών αρχών για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Ισχύει αυτό ή πρέπει να ακολουθήσουμε την παλιά παραδοσιακή μέθοδο. Παράδειγμα, ε, μιλούμε για το darknet, αυτή η συζήτηση γίνεται συνεχώς, πώς θα ε, μπορούμε να διώκουμε εκεί το έγκλημα και έχουμε παραδείγματα αντίστοιχα. Η αστυνομία λοιπόν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον Darknet, δηλαδή οι ίδιοι αστυνομικοί να δημιουργούν λογαριασμούς, να μπαίνουν σε αυτό το σκοτεινό δίκτυο. Η κυρία Χέλγκα Στέβενς από την ομάδα της ΕΣΙΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, Μας είπατε ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της διακίνησης ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών. Επίσης, έχει αυξηθεί σημαντικά ε, ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που εμπλέκονται και μάλιστα είναι και στο στόχαστρο αυτών των διακινητών και των δικτύων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Ρέιν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται λόγος για τους ανηλίκους που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτούς τους καταγράφουμε με βιομετρικά στοιχεία από την ηλικία των 16 ετών και άνω. Αυτό μπορεί να βοηθήσει για να τους προστατεύουμε από τους διακινητές, διότι τα βιομετρικά στοιχεία δεν είναι εύκολο να πλαστογραφηθούν. Ε, συμφωνείτε εσείς με αυτή την άποψη. Και η δεύτερη ερώτηση, πάντα για τη διακίνηση ανθρώπων. Οι διακινητές συνήθω δεν είναι κάτι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε περίπτωση που καταφέρουμε, ας πούμε, να τους συναμβάνουμε, τις περισσότερες φορές αυτή είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης ε, είναι ένα γρανάζι μόνο σε μια ολόκληρη μηχανή. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτό το πραγματικά διεθνές και οργανωμένο έγκλημα για να ανοιχνεύουμε ας πούμε τις οδούς ε, διακίνησης. Μπορείτε να μου απαντήσετε σας παρακαλώ και στις δύο ερωτήσεις, ιδιαίτερα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Είναι πρόθυμες να συνεργάζονται χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Μπέκ από τους Ελεύθερους. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, δύο ερωτήσει πολύ γρήγορα. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά αναλυτική και εις βάθος παρουσίαση αλλά και για την διαπίστωση ότι δηλαδή τα κυκλώματα ενισχύονται χάρη στις έρευνες της Europol που τα εντοπίζει. Ε, θα ήθελα και εγώ πως ε, η συνάδελφος να ρωτήσω το εξή. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τις πρακτικές από χώρα σε χώρα και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ερευνών πόσες περιπτώσεις διλευκάνονται και πόσες συνεχόμενως εγκαταλείπονται ή αρχιοθετούνται. Και δεύτερη ερώτηση. Βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε στους σχετικούς ε, πίνακες όσον αφορά τις ε, συλλαγές που γίνονται στο σκοτεινό ίντερνετ η δουλειά αυτή είναι φυσικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και υψηλής αξίας αν θέλει κανείς δηλαδή να παρακολουθήσει το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, τα δίκτυα παιδοφιλίας ε, και τα άλλα εγκληματικά δίκτυα. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί, πράγμα το οποίο με οδηγεί στην τρίτη παρατήρηση. Βάσει του νέου κανονισμού, τη νέα συντολή, αν θέλετε, τη Europol, που θα αρχίσει να ισχύει σε λίγε μέρε, ε, θεωρείται ότι το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται, αντικατοπτρίζει την σημερινή κατάσταση έτσι όπως την αποτυπώσατε στη μελέτη ή χρειάζονται να προσθήκε κλπ. Πρώτα, πολύ ωραία. Ξεκινούμε τη συζήτηση. Ο Καρλός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βουενράιτ. Λέω κύριο Σκόλιο, όσον αφορά την απάτη στο πλαίσιο του SIS, του Συστήματος Πληροφοριών Σέγγεν. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια, τουλάχιστον 15 χρόνια, έκρεμει μια απάντηση ευρωπαϊκή για την παραχαραξή των εγγράφων. Είναι μια αρμοδιότητα η οποία παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Σύμφωνα με την έκθεσή σας, η παραχαραξή εγγράφων είναι παραγόν κλειδί που διευκολύνει το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και το εμπόριο Ας πούμε, ξέρετε τις υποψίες που υπάρχουν ε, για την επίθεση του Βερολίνο, τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούσαν, όπως εσείς είπατε, πλαστές ταυτότητες. Και λέτε επίσης ότι η χρήση ενισίων διαβατηρίων από τους τρομοκράτες αποτελεί πάλι η βασική μέθοδο εργασία. Όπως γνωρίζουμε στο SAS υπάρχουν 55 εκατομμύρια έγγραφα ταυτότητες, διαβατήρια κλπ. και να τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τον ρόλο που διαδραματίζει το SIS ως οργανισμός ε, στον τομέα αυτών και επιπλέον Τώρα που αλλάζει η νομική βάση, ένα σχόλιο θα ήθελα όσον αφορά τις κείμενες προτάσεις. Έχετε κάποια πρόταση για να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, πιο αποτελεσματικά το SIS για να προλαμβάνουμε ακόμη περισσότερες απάτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Ίσως είμαι εκτός θέματος, αλλά Διάβασα γερμανικέ εφημερίδες την περσμένη εβδομάδα και διάβασα για την γερμανική υπηρεσία, την BND, η οποία κατασκόπευε υποτίθεται την Europol, την Interpol για χρόνια και χρόνια. Παρακολουθούσε τηλεφωνικέ συνομιλίες, ε, email και πολλά άλλα. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, διερευνάται και υπάρχει τρόπο να προστατευθεί η Europol μπορείτε να προστατεύσετε τα στοιχεία σας, τα δεδομένα σας κατά τέτοιων παραδιάσεων. Γιατί αν μια γερμανική υπηρεσία είναι σε θέση να σας κατασκοπεύει, τότε ε, ίσως και κάποιοι άλλοι με ακόμα χειρότερες προθέσεις θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο. Ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτό παρακαλώ. Πρώτα ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Wainwright και πάλι για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω με τη σειρά κυρία Ματσολά. Για τη διαφθορά. Βεβαίως, ανέκαθεν αναγνωρίζαμε ότι είναι παράγον κλειδί για την εγκληματικότητα και το λέμε στην έκθεσή μας. Παραμένει λοιπόν προτεραιότητά μας η διαφθορά. Η συμμετοχή κατά περίπτωση σε υποθέσει, ε, εξαρτάται από του όρου τη εντολή μα. Εμεί δεν μπορούμε να δρομολογήσουμε ανεξάρτητες έρευνε. Οπότε από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σχολιάσω τη μία την άλλη συγκεκριμένη υπόθεση. Εξαρτώμεθα, επαναλαμβάνω, από τα κράτη-μέλη, τα οποία ενδέχεται να μα ζητήσουν να συμμετάσχουμε σε μία έρευνα. Η εντολή μας μας περιορίζει σε περιπτώσεις διασυνοριακές που αφορούν πάνω από δύο κράτη-μέλη και με την προπόθεση ότι καλούμεθα από κάποιο κράτο μέλος. Θεωρητικά ένα κράτο μέλος δύναται να μα καλέσει να διερευνήσουμε ένα έγκλημα, ένα δίκημα σε άλλη χώρα, αλλά αυτό ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο θα έλεγα. Οπότε, εν κατακλείδη, εξαρτώμεθα από το κράτος μέλος, το οποίο υποτίθεται ότι έχουν τελεστεί αδικήματα, τότε καλούμεθα ενδεχομένω να συμμετάσχουμε στις έρευνε. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα της Σίπελ. Όντως, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το πώς επηρεάζει το έγκλημα την κοινωνία. Αυτό το οποίο καταγράψαμε είναι βεβαίως οι οκτώ προτεραιότητες που αφορούν όλα τα κράτη-μέλη σε διαφορετικούς φυσικά βαθμούς όμως εν γέννη για την Ευρώπη στο σύνολό της οι οκτώ τα 8 δικήματα που καταγράψαμε, οι 8 δραστηριότητε είναι κοινέ, κοινού ενδιαφέροντο. Μετά από την έκθεση στο Συμβούλιο, η συζήτηση οδήγησε στην έκφραση ανησυχιών από κάποια μέλη που είπαν ότι ίσως και άλλες προτεραιότητες θα έπρεπε να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, φόρος ε, ΦΠΑ, φόρων κατανάλωση, περιβαλλοντικό έγκλημα κλπ. Έχει δρομολογηθεί αυτή η σχετική συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο και θα κορυφωθεί στις αποφάσεις, ή με τις αποφάσεις των Υπουργών φέτος τον προσεχή Ιούνιο. Και όντω κάποιες κυβερνήσεις ζητούν από τις αστυνομίες τους να αλλάξουν τις τακτικές τους, τις πρακτικές τους. Ξέρετε, χρειάζεται εκπαίδευση, ας πούμε, σε ψηφιακές τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να επαφιέμεθα συνεχώς σε μια πολύ μικρή ομάδα ειδικών. Τώρα πλέον κάθε δίκημα, κάθε έγκλημα έχει πτυχές που αφορούν την πληροφορική. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλοεκπαιδευμένους επιθεωρητές, διερευνητές σε θέματα οι οποίοι έχουν εκπαίδευση και σε θέματα τεχνολογίας. Οπότε αυτό το ζητάμε από τις αστυνομίε μας, ζητάμε περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό κάνει και η Europol και είναι το σημείο επαφή ε, κάθε φορά που μια διερεύνηση, κάθε φορά που μια έρευνα ε, είναι διασυνοριακή. Για το σκοτεινό ίντερνετ, όπω το λέμε, ε, κοιτάξτε, είναι μια τάση δεδομένη αλλά δεν συμβαίνουν τα πάντα εκεί μόνο, συμβαίνουν και στο γνωστό, στο ορατό ίντερνετ αν θέλετε, που παρέχει εχέγγυα ανωνυμίας. Στο darknet, στο ορατό ίντερνετ, και εκεί όμως έχουμε δυνατότητες ε, παρακολούθησης διαφορών δραστηριοτήτων. Αυτό εξαρτάται από την νομοθεσία του κάθε κρατούς μέλους. Η αστυνομία φυσικά έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και στο αόρατο ίντερνετ για να παρακολουθήσει τη μία την άλλη δραστηριότητα. Το πρώτο πρόβλημα βεβαίω, το βασικό πρόβλημα είναι λόγω της κρυπτογράφησης να εντοπίσουμε τους εγκληματίες. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Εδώ πρέπει να βελτιωθούμε. Δηλαδή οι αναλυτικές μας ερευνητικές δυνατότητες στο διαδίκτυο πρέπει να βελτιωθούν, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία στο έπακρο και αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. Όμως η σχετική συζήτηση είναι ακόμη εν εξελίξη. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε όσον αφορά τον διαδίκτυο, πολλά ε, ζητήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Και επίσης για τα βιομετρικά, τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων για άτομα κατά των 8 ή των 6 ετών. Ναι, θα μας βοηθούσε, είναι αλήθεια. Θα μας βοηθούσε να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά και τους ασυνοδευτούς ανήλικους. Σήμερα δεν έχουμε τα σχετικά μέσα όμως, πρέπει να σας πω. Ε, τα βιομετρικά στοιχεία δεν είναι η μόνη λύση. Υπάρχουν και άλλα ενδιάμεσα προσωρινά μέτρα τα οποία μπορούμε να δρομολογήσουμε για να ξέρουμε ποιο μπαίνει και ποιο βγαίνει και, και ιδιαίτερα ε, τι γίνεται με του πιο ευάλωτους πληθυσμού, με τι πιο ευάλωτες ομάδε πληθυσμού. Τώρα για του ε, δουλεμπόρους που είπατε ότι είναι εκτό Ευρώπη όχι πολλοί είναι στην Ευρώπη, έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εντός, εκτός ή και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στον τομέα αυτών της καταπολέμησης του δουλεμπορίου. Πιάσαμε και μεγάλα ψάρια, όχι μόνο τη Μαρίδα. Πάντως το πρόβλημα αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό ξεκινά εκτός Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Η πρόσφατη δήλωση πάντως δίνει την ευθύνη στην Europol να αξιοποιήσει τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι χώρες ε, μέλη, οι χώρες της περιοχής, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του πού βρίσκονται αυτά τα δίκτυα και πώς λειτουργούν, πώς επιχειρούν. Κύριε Κρισπέκ επίσης ρώτησε, ο κανονισμός, ο νέος κανονισμός θα βοηθήσει. Ναι, διότι μας δίνει περισσότερες δυνατότητες, μας λύνει τα χέρια να συνεργαστούμε με τον χώρο της οικονομίας, της τεχνολογίας, κυρίως με τον χώρο της τεχνολογίας, με ιδιωτικές εταιρείε που μπορούν να μας βοηθήσουν. Και σίγουρα θα μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας αντιμετώπισης του εγκλήματος σε μια εποχή που είναι εποχή τεχνολογίας. Επίσης θα βελτιώσουμε την κρατότητά μας να κάνουμε συμπίληση πολύ μεγαλύτερου όγκου δεδομένων να τα αναλύουμε. Στα πλαίσια του κανονισμού λοιπόν θα βελτιώσουμε αυτές τις δυνατότητες. Ε, αυτό είναι και το κυριότερο στοιχείο του νέου κανονισμού. Θα μας επιτραπεί λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορική με πιο έξυπνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικότερες απειλές. Μια άλλη πτυχή της νέας νομοθεσίας είναι ότι βελτιώνει τις μεθόδους διακυβέρνησης και βεβαίως δίνει στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν ε, σημαντικότερο ρόλο επίβλεψης και παρακολούθησης. Κάτι το οποίο είναι νομίζω κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενο από το κοινό. Κ. ρώτησε τι γίνεται με την μεταρρύθμιση του SIS, του συστήματος πληροφοριών Schengen και αν μπορεί να βελτιωθεί. Ε, και τι γίνεται επίση με την παραχάραξη εγγράφων. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Από όλα όσα ανέφερα, ο αυτό, σε αυτή η δραστηριότητα διονγκώνεται ταχύτερα από κάθε άλλον. Δηλαδή, το οργανωμένο έγκλημα έχει ρίξει εκεί το βάρος του. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Ίσως η Europol θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στο σύστημα SIS. Θα μα βοηθούσε. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η ερώτησή είναι ε, εξαιρετικά επίκαιρη και θα επανέλθω αν έχω να καταθέσω περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ πάντως που θέσατε το ζήτημα. Και τέλο, τον κύριο Λένα, σχετικά με του ισχυρισμού τις υπόνοιες ότι μας κατασκόπευε η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν έχω τέτοια στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυτή τη θέση. Συνεργαζόμαστε, όπω φαντάζεστε, με τι γερμανικέ αρχέ βεβαίω. Όμω, να ξέρετε ότι τα μέτρα προστασίας ε, στον τομέα της πληροφορικής, της Europol, είναι εξαιρετικά ε, ικανά και το βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες. Οπότε έχω την πεποίθηση, έχω τη σιγουριά ότι είμαστε καλά, αν θέλετε, από πλευρά προστασία στοιχείων. Δεν μπορώ να αποκλείσω 100% βεβαίω την πιθανότητα ε, κάποιος τρίτος να παρέμβει, αλλά Όσον αφορά τι υπόνοιε ε, κατασκοπία, πραγματικά δεν έχω κάποιο στοιχείο το οποίο να τεκμηριώνει μια τέτοια υπόθεση. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ. Κύριε Γουέντρα, πολύ συγκεκριμένε οι απαντήσει σα και πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Πάρα πολύ χρήσιμη για τα μέλη τη Επιτροπή και προχωρούμε στο σημείο υπαριθμών έρεξη στην ημερήσια διάταξη. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψε με ειδικού σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Ε, as a reminder, this exchange of views is organized... Όπως σας θυμίσα, αυτό γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας που ζήτησε η Επιτροπή μας για το ίδιο θέμα έχετε λάβει ένα χωριστό πρόγραμμα με τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων που έχουμε προσκαλέσει και σύντομη παρουσίαση των οργανώσεων και των οργανισμών που εκπροσωπούν. Το πρώτο τμήμα της ε, συνεδρίασης θα διαρκέσει μία ώρα περίπου και θα έχουμε τις παρουσιάσεις των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων ε, που καλέσαμε βάσει της απόφασης των συντονιστών. Μάλιστα. Αρχίζουμε με τις παρουσιάσεις των προσώπων think tank της κοινωνίας των πολιτών και γενικότερα για το hacking και μετά θα ακολουθήσουμε την Eurojust και τη Γενική Διεύθυνση Home, τη Γενική Διεύθυνση Just. 45 λεπτά θα είναι το δεύτερο τμήμα της ακρόασης με ρωτήσεις και απαντήσεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή και στους κοιόδης για την καταπολέμηση των κλίματος στον κυβερνό χώρο. Και άμα το επιτρέψει ο χρόνος, θα ακούσουμε και άλλα μέλη. Πρώτα όμως οι εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει. Πραγματικά σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Πέντε λεπτά ο καθένας. Ο ε, ε, πρώτος, ο κύριος Μπεχτράν Λασαπέλ, εκτελεστικός διευθυντής ε, Ιντερνετ και Jurisdiction. Thank you very much. Um, for the opportunity to... Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνω αυτή την παρουσία στην Επιτροπή. First, uh, let me... Επειδή έχω το προνόμιο να μιλώ πρώτος, θα ήθελα να σας θέσω ίσως στο γενικότερο πλαίσιο ε, τη δικαιοδοσία στην καταπολέμηση του κλίματος του κυβερνοχώρου κάπως ευρύτερα και όχι με τη στενή έννοια δηλαδή του ηλεκτρονικού εγκλήματος διότι τα προβλήματα δικαιοδοσία στην καταπολέμηση των καταχρήσεων ε, διαπερνούν ε, πολλά θέματα. Δεν θα κάνω ένα εξαντλητικό κατάλογο, αλλά έχουμε τεχνικές καταχρήσεις, το phishing, τα ε, λογισμικά, τα ε, κακόβουλα κλπ. Και επίσης ε, διάδοση περιεχομένου που μπορεί να είναι νόμιμο σε μια χώρα αλλά παράνομο σε μια άλλη χώρα, παρενόχληση, συγκοφαντική δυσφήμιση, προώθηση εξύπριση της τρομοκρατίας κτλ. Αλλά αυτό συνδέεται και με δραστηριότητες uh, που μπορούν να είναι λαθρεμπόριο ε, προϊόντων ε, στο διαδίκτυο, όπως είναι πλαστά φάρμακα ή πλαστά προϊόντα. Ε, εγώ θέλω να ασχοληθώ λοιπόν σήμερα με τα προβλήματα για τη δικαιοδοσία για την κάλυψη αυτών των αδικημάτων. Τα έφερε και ο κύριος Γουέν Ράιτ, υπενήχθη. Είναι ένα ευρύ φάσμα λοιπόν αυτό, το οποίο εξετάζουμε. Ποιε είναι οι προκλήσεις. Τρία στοιχεία είναι πνές, αλλά αξίζει να το επαναλάβουμε ότι το διαδίκτυο και οι υπηρεσίε που παρέχει είναι διεθνείς και προφανώς το οργανωμένο έγκλημα και το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι διεθνές. Για παράδειγμα, οι εταιρείε ε, αποθηκεύουν κάποια στοιχεία για τους πελάτες τους, για τους χρήστες. Ε, και αυτό μπορεί να καλύπτεται από διαφορετικές δικαιοδοσίες και επίσης η πρόσβαση των προφοριών είναι διαφορετική. Αυτό Μα έτσι αντιμέτωπους με πολλά προβλήματα και προβλήματα επιβολής ε, τη εθνική νομοθεσία και προβλήματα ορισμού ή εντοπισμού για το ποιο δίκαιο εφαρμόζεται με την κλασική παραδοσιακή έννοια. Δεν είναι εύκολο πάντα αυτό να υλοποιείται στο διαδίκτυο. Και όταν η παρανομία είναι διεθνής, Μπορεί μάλλον να είναι διεθνής η παρανομία, αλλά η η ένωμη τάξη κάθε χώρα είναι ε, κάτι που αφορά την επικράτειά της και τίθεται ζητήματα κυριαρχίας. Ακόμα αν το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί οι περισσότεροι ευρωπαίοι χρήστε χρησιμοποιούν υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες περιφέρειες εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Άρα τίθεται το θέμα εδώ της ετεροδικία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, της ε, Αν μιλήσετε με προσώπους ε, της αστυνομίας ή και των εταιριών που αντιμετωπίζουν τέτοιες παρανομίες, ποια είναι η ηρωνία που θα διαπιστώσετε. Όλα τα συστήματά μας βασίζονται σε κάποια δικαιοδοσία εθνική, κρατική, σε μια επικράτεια, η οποία σήμερα αντί για λύση έχει καταστεί πρόβλημα, γιατί χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία και τα διεθνή εργαλεία συνεργασίας δυστυχώς δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένα. Θα επεκταθώ. Αν ξέρετε το ε, σύστημα για ε, τις συμφωνίες και τις συμβάσεις αμοιβαία δικαστικής συνδρομής, βλέπω να με διάτε, ε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να εφαρμόζεται κάθε φορά και να χρησιμοποιείται αυτή η διαδικασία. Επειδή πιέζει ο χρόνος, θέλω να τονίσω το εξή. Αυτό το θέμα της δικαιοδοσίας κάθε κράτους στην επικράτειά του πρέπει να λυθεί και γίνονται προσπάθειες ε, να λυθεί κυρίω για την πρόσβαση σε δεδομένα που αποθηκεύουν κάποιες εταιρείε. Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από το γεγονός και μόνο, ας πούμε, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πολλές φορές κάποιες εταιρείε που εδρεύουν στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν νομικά προβλήματα. Όταν κάποιος του ζητάει να δώσουν πληροφορίες για τους χρήστες στα πλαίσια μιας διερεύνησης ενός εγκλήματος, είναι υποχρεωμένες να επιλέξουν ποιο δίκαιο θα παραβιάσουν. Διότι υπάρχει η νομοθεσία για το ιδιωτικό των ε, συνομιλιών και των επικοινωνιών ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχεται σε αντίφαση με αυτά που ζητούν τα κράτη-μέλη μας. Ε, γίνονται πολλά αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες για να ε, προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και ένα από τα μεγάλα θέματα που θέλω να σας αναφέρω είναι η συνεκτική πολιτική και η συμβατότητα. Ένα άλλο στοιχείο που έχει σημασία είναι να αναγνωρίσουμε το ρόλο των ιδιωτών φορέων εδώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις Εκείνοι που καταχρώνται ή παρανομούν στο διαδίκτυο το κάνουν με στοιχεία που έχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που αποθηκεύουν ε, τα στοιχεία αυτά και οι δραστηριότητες πολλές φορές μπορεί να είναι νόμιμες σε μια χώρα και παράνομες σε μια άλλη. Ε, πολλές φορές λοιπόν αυτοί οι πάροχοι ε, υπηρεσιών διαδικτύου ή μεσολαβητές ε, έχουν σημασία γιατί συμμετέχουν στον ορισμό των κανόνων. Σήμερα οι εταιρείε ε, καμιά φορά έχουν λόγο για το τι μπορεί να κάνει ένας χρήστης, τι μπορεί να αναρτήσει ή να μην αναρτήσει ε, σε αυτό το χώρο που λέγεται κυβερνοχώρος και αυτό αφορά εκατομμύρια χρηστών. Ένα άλλο στοιχείο που καθιστά τι εταιρείε πολύ σημαντικές είναι ότι σε κάποιο βαθμό έχουν τη δυνατότητα επιβολή κιόλας του νόμου, διότι μπορούν να ε, διακόψουν ένα λογαριασμό, να αφαιρέσουν περιεχόμενο ή να το φιλτράρουν. Άρα, όταν ε, μιλούμε για τους κανόνες και ποιους ε, ισχύουν, ε, που ισχύουν, για ποιους ισχύουν και ποιος τους επιβάλλει, αυτό πολλές φορές είναι στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Και πολύ σοβαρότερο είναι ότι πολλές φορές αυτές οι εταιρείες δεν έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το τονίζω αυτό, διότι στη συζήτηση ε, περί καταπολέμησης εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και καταχρήσεων γενικά, αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τα κράτη-μέλη, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο και οι ιδιωτικές εταιρείες οι οφείλουν να διαδραματίσουν. Και τέλος, σε σχέση με τις γενικότερες προκλήσεις και προβλήματα που έχουμε, θα πρέπει να ξαναδούμε ε, ε, μάλλον να ε, συμφιλιώσουμε αντικρουόμενους στόχους. Δηλαδή να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, σεβόμενοι όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και διασυνοριακά. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον εντάσεων λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του διαδικτύου, ενώ είναι εθνικός, επαναλαμβάνω, ο χαρακτήρας της νομοθεσίας, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Υπάρχει μια φυσική τάση που είναι πάρα πολύ κατανοητή να χρησιμοποιούμε την κείμενη νομοθεσία, τα εργαλεία που διαθέτουμε, την εθνική νομοθεσία προκειμένου για διεθνείς συμφωνίες. Το πρόβλημα όμω ποιο είναι. Επειδή έχουμε ένα αίσθημα, τα κράτη συγκεκριμένα, ε, ότι είναι ανήμπορα απέναντι σε αυτές τις ε, καταχρήσεις, τείνουν να υπερβάλλουν. Θα σας αναφέρω μερικά στοιχεία προτείνουν ως λύση την υποχρεωτική ε, ανείχνευση και τον εντοπισμό των στοιχείων. Αυτό τεχνικά δεν γίνεται πάντα. Και ε, ενδέχεται να είναι εις βάρος και αναπτυσσόμενων μικρών εταιρεών και αναπτυσσόμενων κρατών. Θα επανέλθω αργότερα σε αυτό αν θέλετε στη συζήτηση. Μια δεύτερη τάση που παρατηρούμε είναι να επεκταθεί ε, η ε, δικαιοδοσία ε, του κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της επικράτησης και να χρησιμοποιεί δηλαδή το κράτος στην ετεροδικία. Αυτό και πάλι χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό και ε, λελογισμένη χρήση, γιατί μπορεί κάποιες εθνικές ή ε, περιφερειακές αποφάσεις να έχουν επιπτώσεις και ισχύ για ε, φορείς εκτός της επικράτειας. Και αυτό μπορεί να είναι μια κούρσα νομικών όπλων, ας πούμε, που μπορεί να είναι επικίνδυνη. Τρίτον, η χρήση κάποιων ενδιαμέσων, μεσαζόντων. Υπάρχει ένας η χρηση καποιων ενδιαμεσων ζωντων εδώ να ρίξουμε όλη την ευθύνη στις εταιρείε που τελικά θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για το ποιο νόμο θα χρησιμοποιήσουν ή ποιο νόμο θα παραβούν. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς ε, σωστή διαδικασία. Και αυτό είναι επιπλέον εμπόδιο ε, ε, για τις εταιρείε αυτές και βάρος. Και τέταρτο το Domain Name System ε, μπορεί ε, να χρησιμοποιηθεί για να λυθούν κάποια ζητήματα. Αλλά εδώ χρειάζεται και πάλι προσεκτικός χειρισμός. Γιατί οτιδήποτε κάνει και ε, κάποιος έχει παγκόσμια εμβέλεια. Οπότε θα πρέπει να είναι και κάπω ε, παγκόσμια η παρανομία ή το έγκλημα για να δικαιολογείται παγκόσμια δράση. Συμπέρασμα. Σε αυτό το περιβάλλον ε, υπάρχει έντονη ανάγκη συνεργασίας των ε, ενδιαφερομένων, των εμπλεκομένων, σε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Και χρειάζεται ένας χώρος για να συζητούν αυτοί οι φορείς. Γι' αυτό και εμείς από το 2012 στο Internet και Jurisdiction που είναι ένα δίκτυο ε, όπου συγκεντρώνονται πάνω από 200 ενδιαφερόμενοι, ιδιώτες, τεχνικοί, φορείς, κοινωνία των πολιτών, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστημιακοί έχει τρία προγράμματα. Το πρώτο αφορά τα δεδομένα και τη δικαιοδοσία για τις διασυνεργειακές ε, διώξεις και έρευνες. Το, δεύτερο έχει να κάνει με το περιεχόμενο και τη δικαιοδοσία και πώς αφαιρείται αυτό. Και το τελευταίο αφορά το DNS ε, και πώς διακόπτεται η σύνδεση ενός ενώματος μία Επειδή τελειώνει, τελείωσε ο χρόνος μου, πέρσι τον Νοέμβριο κάναμε την πρώτη μας διάσκεψη ε, που συγκεντρώθηκαν 200 φορείς με τρεις ομάδες εργασίας ή ομάδες επαφών για το κάθε θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον εκτελεστικό ε, σύμβουλο του Defending Rights and Freedom Online, τον κύριο Μακνάμι. Το όνομα της οργάνωσης είναι τα Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και τους εισηγητές. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω τον ρόλο των μεσαζόντων πολλές φορές είναι πολύ εύκολο να ε, υπάρχει περιορισμός ε, της δράσης συγκεκριμένων φορέων έτσι ώστε να μην μπορέσουν να δράσουν ελεύθερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ε, ορίσει την δράση των μεσαζόντων με βάση των, τις διάφορες οδηγίες ως προσοκόπηρα, η τρομοκρατία, τη ρητορική μίσους και την ε, οδηγία που αφορά την ε, χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Και θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μία οριζόντια προσέγγιση με βάση αποδεικτικά στοιχεία και την πείρα μας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μία ομάδα εμπειρογνωμών που ασχολείται με το ρόλο των ε, μεσαζόντων και που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να κατανοήσουμε αυτόν τον τομέα πολιτικής μας. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία σε σχέση με την μελέτη που προετοιμάστηκε για την Επιτροπή αυτή. Το, την προσέγγιση «Going Dark» και το πώς μπορούμε να δράσουμε έτσι ώστε να, αντιμετωπί... να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη... τα διάφορα λογισμικά hacking. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρησιμοποιούμε την έννοια της χρήσης του σκοτεινού διαδικτύου, going dark, και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αποδυναμώσουμε τα συστήματα κρυπτογράφησης. Πρόκειται για έναν όρο ο οποίος μπορεί να ε, οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Αυτός ο όρος going dark. Στην πραγματικότητα Ζούμε στην χρυσή εποχή εποπτείας και υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο εποπτείας. Υπάρχει γεωπροσδιορισμός, ε, στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνικές διαδράσεις μέσω του like, dislike, κάτι το οποίο δεν υπήρχε 20 χρόνια πριν. Άρα μπορούμε να ε, δούμε κατά πόσο μπορεί να αποθυναμωθεί η κρυπτογράφηση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που δεν υπήρχαν 20 χρόνια πριν. Έγινε μνήα και σε μία ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας. Τη στιγμή που υπάρχει κοινωνική διάδροση επιχειρηματική και διακυβερνητική, δεν θα πρέπει να θεωρούμε τον κυβερνοχώρο σαν κάτι το αφηρημένο. Υπάρχει λοιπόν ασφάλεια γενικότερα, όχι κυβερνοασφάλεια. Μιλάμε για μία σχέση κόστους-οφελίας. Δεν μιλάμε για ασφάλεια έναντι κυβερνοασφάλειας. Μιλάμε για ασφάλεια σε σχέση με τις ελευθερίες. Όταν μιλάμε για hacking από τις δημόσιες αρχές, θα πρέπει να δούμε τη σχέση κέρδους, ε, ωφελίας μάλλον, και ζημίας. Σε σχέση δηλαδή με τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να ορίσουμε τις ευαλωτότητες που ε, υφέρπουν και δεν θα πρέπει να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σε όλους τους χρήστες του συστήματος. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για αυτά τα είδη ευαλωτότητας έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το έγκλημα και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δίκτυα εγκληματικές οργανώσεις μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης ευαλωτότητας του συστήματος πιστεύω ότι αυτές οι ευαλωτότητες ε, γίνονται πιο επικερδείς γιατί ο κύριος ε, Wainwright μίλησε για το έγκλημα ως υπηρεσία. Πολύ σωστά μιλάμε για έναν κίνδυνο έλλειψης ασφαλείας ε, ως προς τη χρήση του συστήματος από δημόσιους φορείς θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε ε, το σύστημα έτσι ώστε οι εταιρείες λογισμικού να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διασυνοριακή πρόσβαση σε στοιχεία απόρριτα ή μη. Η DG Home και DG Just έχουν προβεί σε ενδελεχή εργασία σε αυτό το τομέα, την οποία, προς, την οποία ε, προσετεριζόμαστε. Έχω υπερβεί το χρόνο μου, το ξέρω, η Europol όμως θα κατάφερε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή κατάφερε να σπάσει δύο κωδικούς κρυπτογράφησης σε σχέση με ένα δίκτυο ε, Η Λούση Κραχούλσοβα από, την ε, Ευρωπαϊκή, από πλευράς Ευρωπαϊκής Πολιτικής ε, Συνδρομής. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους βουλευτές της Επιτροπής που επικοινωνούν με τους αρμόδιους φορείς. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Λούση και εργάζομαι για Διεθνή ΜΚΟ υπέρ των ε, ψηφιακών δικαιωμάτων σε ολόκληρον τον κόσμο. Με βάση την εμπειρία μας, το διαδικτύο είναι ένας κατεξοχήν χώρος για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υποστηρίζουμε έτσι την τεχνολογία, την πρόοδο και την πρόσβαση σε αυτά. Εξασφαλίζουμε περισσότερη διαφάνεια, αποκλεισμένοι άνθρωποι επικοινωνούν, οι καλλιτέχνες δημιουργούν, οι ερευνητέ ερευνούν και η πρόοδος αφορά και πολλούς άλλους ε, τομείς όπως η ε, υγεία. Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική υποδομή υπέροχη από την ε, μία μεριά, όπως προανέφερα, με κινδύνους όμως από την άλλη, κάτι το οποίο οδηγεί σε περισσότερη νομοθεσία για την προστασία των χρηστών, καμιά φορά και σε υπονόμευση της λειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει λοιπόν από την άλλη μεριά ότι οι νομοθέτες ε, βλέπουν το διαδίκτυο ως πιθανό στόχο από εγκληματίες με προηγμένη τεχνολογία. Καμιά αυτό αφορά και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Από την άποψη λοιπόν των ε, κοινωνιών μας βλέπουμε το διαδίκτυο να χρησιμοποιείται και ως όπλο. Μέσω του διαδικτύου επίσης ασκούμε παρακολούθηση και αυτό είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο, δηλαδή κυβερνήσεις και οι αστυνομίε ε, βλέπουν να εξωθούν στα όρια του σχετικού κανόνες εκμεταλλευόμενες τα, την τροτόρυτα των επικοινωνιών. Γι' αυτό η μάχη που δίνουμε στο διαδίκτυο είναι δύσκολο να κερδιθεί. Ο έλεγχος του διαδικτύου είναι απολύτως αδύνατος. Φυσικά οι επιτιθέμενοι έχουν το πλεονέκτημα, έχουν το πάνω χέρι. Το μόνο που χρειάζονται είναι μια μικρή τροτότητα εντοπισμένη για να δράσουν. Και αυτό θέτει το θέμα της προστασίας του διαδικτύου. Τα πιθανά σενάρια είναι πάμπολα. Κινδυνεύουμε όλοι στο σπίτι μας, στην κρυβατοκαμαρά μας, κινδυνεύουμε τα παιδιά μας, οπότε το θέμα είναι να καθορίσουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Πού βρίσκονται τα όρια διάφορες ε, κακόβουλες ε, συσκευές και λογισμικό πλήττουν καθημερινά τις τιμέ. Αυτό αφορά όλους τους χρήστες, τους καθημερινούς απλούς χρήστες. Οι νομοθέτες λοιπόν πρέπει να μας προστατεύσουν χωρίς όμως να υπονομεύουν τα δικαιώματά μας. Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Εμείς από την πλευρά μας, την πρόσφατη έκθεσή μας σχετικά με το hacking των κυβερνήσεων υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στην έκθεση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η βάση των απειλών κατά της ιδιωτικότητας και της ελεύθερης έκφρασης καθώς και τη στήριξη των κανόνων πολιτικής δικονομίας πρέπει να ληφθούν απαραίτητα μέτρα. Το κοινό ζητά περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τους ε, κανόνες που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις για το hacking. Θέλουν οι κανόνες δικονομίας να εφαρμόζονται και θέλουν διαφάνεια όχι για τη διαφάνεια, αλλά επί της ουσίας. Το hacking αποτελεί σίγουρα απειλή για τις επικοινωνίες και τις συσκευές μας. Τέλος, προτείνουμε 10 κατευθυντήριες γραμμέ προστασίας κατά του hacking των αρχών και των κυβερνήσεων. Θα παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και την σχετική έκθεση για το κυβερνητικό hacking, όμως να σας, για να σας προειδεάσω, αυτό το οποίο βασικά λέμε είναι ότι πρέπει πρώτον αυτό το hacking να προβλέπεται από νόμο, για να μην στιγματιστεί το κυβερνητικό χάκι χωρίς λόγο. Επίσης, τα μέσα πρέπει να είναι τα λιγότερο επιθετικά, θα έλεγα, και να έχουν και περιορισμό στο χρόνο. Ό,τι γίνεται, ότι ισχύει το ή άλλως με τους άλλους κανόνες σχετικά με τις παρακολουθήσει. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που το κράτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κυβερνό έγκλημα. Αυτό πρέπει να γίνει με νομίμους τρόπους, ώστε να όλα αυτά γίνονταν όχι στο διαδίκτυο, αλλά με τους κλασικούς τρόπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο James Eager, ε, σύμβουλο στην Καντάν Λιζέ μάλλον και στον Καντάλιζερ, ε, Επίση σύμβουλο στο ε, Optimity Advisors Europe. Εγώ λέγομαι Quentin και ο συνάδελφος James θα παρουσιάσει τη μελέτη. Έχετε μερικά αντίτυπα εδώ για ε, το νομικό πλαίσιο και τρόπο αντιμετώπισης του hacking. Είναι 50 σελίδες με παραρτήματα που μπορείτε να δείτε και να τα μελετήσετε. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε ένα δεκάλεπτο να τα συνοψίσουμε. Αν θέλετε ερωτήσεις, με χαρά να τις απαντήσουμε ε, στη συνέχεια. Σας είπα, έχουμε μερικά αντίτυπα στην είσοδο της αίθουσας. Μια σύντομη λοιπόν παρουσίαση μου είπα να κάνω τώρα. Ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να σας παρουσιάσω λίγο το πλαίσιο στο οποίο έγινε η μελέτη. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που εξετάσαμε φυσικά το going dark και ζητώ συγγνώμη που ε, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε αυτά. Ε, ποια είναι η υποκείμενη ιδέα. Όσο ε, αυξάνεται η τεχνολογία κρυπτογράφησης ε, που είναι προφανώς απαραίτητη για την ασφάλεια στο διαδικτύο. Αυτό αφορά τα πάντα και τα κινητά τηλέφωνα, τα ATM των τραπεζών, ε, διάφορα συστήματα επίγοντα. Είναι κρίσιμη η κρυπτογράφηση, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει ακριβώς την ε, χρήση από διάφορες χρήσεις πληροφορία με ένα ασφαλή τρόπο ή σε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως τι διαπιστώνουμε. Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν λιγότερη πρόσβαση σε κάποιες από τι πληροφορίε που είχαν στο παρελθόν λόγω της κρυπτογράφησης. Ακούστηκε και προηγουμένω αυτό και μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια θέλετε. Άρα μειώνεται η δυνατότητα των αρχών επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση σε αποδεκτικά στοιχεία και online και offline. Θυμάστε την υπόθεση μεταξύ Apple και FBI για την περίπτωση Σαν Βερντίνο. Ε, τώρα αυτό είναι ένα τμήμα της λύσης, είναι η ίδια η λύση. Είναι η χρήση τεχνολογιών hacking προς όφελος ε, των ερευνητικών σκοπών της αστυνομίας. Να σας εξηγήσω. Γιατί χρησιμοποίησαμε τη λέξη hacking. Φυσικά ήταν και στη μελέτη, αλλά ξέρω ότι οι διαφορετικές αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών όταν λένε hacking ε, ε, εννοούν άλλο τρόπο μάλλον ε, ή κάποιο, κάτι διαφορετικό. Τι κάνουν ουσιαστικά. Ε, έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα ε, ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πληροφορικής, μέσω παρανόμων ας πούμε τρόπων ή όχι πάρα πολύ ορθόδοξα. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ και ποια είναι τα στοιχεία που εξετάσαμε. ασχοληθήκαμε κυρίως ε, με δύο πτυχές του θέματος, η ε, ασφάλεια απέναντι στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ή η ασφάλεια απέναντι στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στο ε, ίντερνετ. Σε αυτό αναφέρθηκαν προσδέσεις με τρόπο πάρα πολύ εκτενή και αναλυτικό. Επίσης, τι συμβαίνει όταν χακάρει η αστυνομία. Θυμάστε τι έγινε με τις κάτω χώρες και τον Καναδά. Ε, είναι η περίπτωση Enet αν δεν απατώμε. Οι ιδιοκτικές αρχές ε, βρήκαν 7 παραμπάιτ, 86 ε, εκατομμύρια σελίδες δηλαδή, καταλαβαίνετε για πόσα στοιχεία και δεδομένα μιλούμε και γιατί όγκο δεδομένων. Περνούμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια σύντομα να σας παρουσιάσω τη μελέτη και την ε, μέθοδο που ακολουθήσαμε. Είδαμε ποια είναι ε, η διεθνή συζήτηση, ε, πού μπορεί να υπάρχει νομική βάση για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι γίνεται με τη συνεργασία διαφορών κρατών μελών. Έξι κράτη-μέλη μελετήσαμε, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, κάτω χώρες, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο και τρεις χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ε, καλές τεχνικές, λιγότερο καλές, πάντως έχουν αναπτυγμένες ε, τεχνικές χακαρίσματος ε, και αυτές είναι η Αυστραλία, το Ισραήλ και οι όπου οι διεκτικές αρχές καταφεύγουν στο hacking. Και επίσης έχουμε και κάποιες συστάσεις και προτάσεις για πολιτική. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω εγώ. Σύντομα να σας πω ποια είναι τα βασικά μας ευρήματα δεν μπορούμε προφανώς να καλύψουμε 50 σελίδες μελέτη σε 10 λεπτά μέσα. Ε, συγκριτική ανάλυση λοιπόν των νομικών πλαισίων των διαφόρων κρατών, έξι κράτη-μέλη στα οποία μελετήσαμε την κατάσταση. Και τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν οι ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ε, τα δικαιώματα, όπως βλέπετε από τη διαφάνεια και τα έξι κράτη-μέλη είναι αυτή τη στιγμή ε, σε διαδικασία έγκρισης ε, δυνατοτήτων ε, χρήσης τεχνικών hacking από την αστυνομία. Το 2016 το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία και έχουν προσαρμόσει το νομικό τους πλαίσιο. Άλλες χώρες το κάνουν αυτό το καιρό από τις 6. Παρ' όλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο ε, που να μπορεί να χρησιμοποιεί η αστυνομία για να χακάρει με την παραδοσιακή κλασική έννοια των διοκτικών αρχών. Παράδειγμα, στη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έχει τη δυνατότητα ε, να το κάνει στα πλαίσια των ε, ποινικών ερευνών. Αλλά γενικά υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στην νομοθεσία σε ε, ό,τι αφορά την παράνομη αυτή η δραστηριότητα τροποντινά των διεκτικών αρχών. Υπάρχει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ο εισηγητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με ε, πολύ σαφείς διατάξεις. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα εργαλεία ε, που χρησιμοποιεί μια διοκτική αρχή, ε, τα επιθετικά κατά κάποιο τρόπο που δεν ταυτίζονται πάντα με το hacking. Εμείς επικεντρωθήκαμε ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, είναι περιορισμένες οι ε, νόμιμες ε, διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Μελετήσαμε τη διαφορά που υπάρχει στις ασφαλιστικές δικλείδες και στη ισορροπία ασφάλειας με ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδη δικαιώματα. Ακούσαμε για τις αποφάσεις δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιορισμοί που έχουν να κάνουν με τη χρονική διάρκεια χρήσης ε, τεχνικών hacking, ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει πρώτερη έγκριση και παρακολούθηση από αρμόδιους οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο. Η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα και υπάρχουν και πολλές επικρίσεις. Παράδειγμα, στην Πολωνία, η Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει μελετήσει ε, σε μεγάλο βάθος τις νέες αυτές διατάξεις. και επικρίνουν και το χρόνο που χρειάζεται για να δοθεί η πρώτερη έγκριση. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία βέλτιστων ή καλών πρακτικών. Σε περίπτωση που θεωρείται απολύτως απαραίτητη η τεχνική αυτή από την αστυνομία, Στη Γερμανία, α πούμε, γίνεται ένα έλεγχο και μετά διαγράφονται κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική ζωή των ενδιαφερμένων. Και στην Ιταλία υπάρχουν κάποια τεχνικά μέτρα που προκρίνονται για την ε, χρήση του hacking. Γενικότερα επιτρέπεται όμως και δεν είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο ή πιο περιοριστικό σε σχέση με άλλες τεχνικές ε, λιγότερο διεισδυτικές. Οι δύο τελευταίες ε, διαφάνειες ε, καλύπτουν τις συστάσεις και τις προτάσεις πολιτικής. Το πρώτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και μετά ακολουθούν οι πολιτικές που προτείνουν. Επειδή όλα αυτά τα θέματα είναι κάπως χαρτογράφητα είδατα ακόμα ε, ως προς τη νομική ε, προστασία και τον έλεγχο και τη βελτίωση των συστημάτων από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα να καταλάβει τι συμβαίνει στην πράξη και μετά ε, τι θα πρέπει, για να προχωρήσει σε συστάσεις, τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει. Θα πρέπει κάθε ε, απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή να λαμβάνει υπόψη ε, τους κινδύνους ε, κάθε φορά που συνδέονται με αυτή και χρειάζεται μελέτη αντικτύπου κάθε φορά από τα κράτη-μέλη πριν προχωρήσουν σε νομοθεσία που να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Χρειάζεται επένδυση σε έρευνα για να κατανοούμε αυτά τα θέματα καθώς προχωράει η τεχνολογία και η χρήση στην πράξη. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία τώρα να ηγηθεί σε όλη προσπάθεια ε, και να συντονίσει την ε, αστυνομία, τη δικαιοσύνη, την κοινωνία των πολιτών, την προστασία των δεδομένων των πολιτών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με τον ε, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη ΣΥΠΟΛ και την Eurojust. Αυτά. Νομίζω ότι συνοψίζουν αυτά τη μελέτη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα βρείτε τα στοιχεία μας ε, εδώ για να αποταθείτε θέλετε να μας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επικεφαλή των ε, επιχειρήσεων αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού εγκλήματος στον ε, κυβερνοχώρο. Ονομάζομαι Φερνάντο Ρουίσε και θα παρουσιάσουμε μαζί με τον συνάδελφο της Eurojust αυτή τη μελέτη. Πρόκειται για ένα κοινό έγγραφο της της Europol και της Eurojust που αφορά τις κοινέ προκλήσεις καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο όλα τα θέματα ε, είναι πολυσχηδή και θα χρειαζόταν ε, κανείς πολύ χρόνο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Σε περιορισμένο χρόνο είναι δύσκολο να έχετε μία σωστή εικόνα. Μπας περιπτώσει θα σας πω ποιες είναι οι προκλήσεις από πλευράς ε, εφαρμογής του, του νόμου. Καταρχήν έχουμε απώλεια στοιχείων, απώλεια δεδομένων. Πολλές φορές ε, δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα. Τα χάνουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι η παρακράτηση στοιχείων. Το 14 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι η αποθήκευση δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν αποθηκεύουν αυτά τα στοιχεία. Ορισμένα κράτη έχουν βεβαίως και θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτά. Η κρυπτογράφηση επίσης είναι ένα περίπλοκο θέμα γιατί πολλές φορές η κρυπτογράφηση έχει διαφορετικές μορφές όταν πρόκειται για κρυπτογράφηση φακέλου ή διαλόγου. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο hardware και ο δικαστής πάντα θα μας πει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία με όλα τα μέσα γιατί ε, αν πρέπει δηλαδή να διαρρήξουμε ένα ε, χρηματοκιβώτιο για να βρούμε τα στοιχεία θα πρέπει να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι όμως όταν δεν έχουμε τεχνικά μέσα για την ε, πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τι κάνουμε. Τότε πάμε στην πηγή, στον, στον κατασκευαστή και του λέμε να μας βοηθήσει. Πολλές φορές μπορεί και άλλες όχι, ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης του λογισμικού. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ή όχι. Αυτή είναι η ουσία της συζήτηση. Σε σχέση με το κρυπτο ε, συνάλλαγμα, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά τα δεδομένα, διότι πολλές φορές γίνονται ε, πληρωμές για εγκληματικές δραστηριότητες και δεν υπάρχει σαφήνεια για το πόσο, πώς μπορούμε να αποδώσουμε τις συναλλαγές σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Γιατί αν έχει γίνει ένα έμβασμα σε μια, από μια συγκεκριμένη πηγή σε κάποιον θα πρέπει να δούμε εάν έχει γίνει και μια συναλλαγή με αλλαγή νομίσματος και πολλές φορές είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί και είναι δύσκολο να μας παράσουν αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, η έλλειψη ε, προσδιορισμού χώρου είναι ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί. Γιατί πολλές φορές οι χρήστες του σκοτεινού διαδικτύου μπορούν να αποθηκεύσουν ένα περιεχόμενο στο διαδίκτυο χωρίς να ξέρουμε πού έχει αποθηκευτεί. Δηλαδή σε ένα εγκληματικό φόρουμ οι εγκληματίες ανταλλάσσουν πληροφορίες για το πώς βιάζουν μικρά παιδιά, αλλά είναι δύσκολο να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Και αν προσφύγετε στη δικαιοσύνη, ο δικαστής θα σας ρωτήσει πού ακριβώς γίνεται αυτό. Αυτοί οι εγκληματίες πού βρίσκονται, δεν ξέρουμε. Επίσης, η πρόσβαση δεδομένων νέφους το θέμα είναι περίπλοκο, διότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν την υπηρεσία μπορεί να μην αποθηκεύουν τα δεδομένα σε μία χώρα, αλλά σε μία τρίτη χώρα. Πάτε λοιπόν στον πάροχο, ζητάτε την ε, πρόσβαση, αλλά δεν μπορεί να χορηγηθεί, γιατί υπάρχει διαχείριση από άλλη χώρα και πολλές φορές τα στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και είναι πολύ δύσκολο να συλλέξετε όλα τα στοιχεία από όλες τις δικαιοδοσίες. Επίσης, ως προς την συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα για ότι έχει μία πολύ καλή θεώρηση της κατάστασης στο χώρο του εγκλήματος. Χρειάζεται βεβαίως μία, ένα νομικό υπόβαθρο, ένα νομικό πλαίσιο και επίσης η θέληση του ιδιωτικού τομέα για συνεργασία, γιατί μπορεί να έχει πληροφορίες, αλλά να μην θέλει να τις δώσει σε τρίτους. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η σωστή νομική πλαισίωση για την ε, επικοινωνία και χορήγηση στοιχείων μέσα στα πλαίσια των κανονισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στη Europol συνεργαζόμαστε με τις αρχές ε, δικαιοσύνης, υπάρχουν συμβουλευτικές ομάδες και έχουμε ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και Εμπιστοσύνη. Γιατί ο ιδιωτικό τομέα δεν είναι υποχρεωμένο να χορηγήσει αυτά τα στοιχεία. Θα κάνει σε θελούσια ε, βάση. Σε σχέση με τη συνέργεια ε, δημόσιο-ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση του, του διαδικτύου Internet of Things. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι στοιχεία ε, χρησιμοποιούμε και ποια, ποια είναι πηγή προσβασιμότητας, ένα smartphone, ε, ένα λάπτοπ και ούτω καθεξής. Και δεν υπάρχει ασφάλεια εξορισμού. Κάθε σύστημα είναι ευάλωτο σε οποιαδήποτε απειλή. Έχουμε πολλά παραδείγματα σε σχέση με την επίθεση του Internet of Things και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με την βιομηχανία για να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας σε όλες αυτές τις συσκευές. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει επί του παρόντος και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Εμείς θίγουμε τα προβλήματα. Η λύση θα έρθει από την ομοθέσια, Θα πρέπει να υπάρχουν ε, ελάχιστες ε, προδιαγραφές ασφάλειας. Ακόμα και όταν πολλούμε ένα παιχνίδι στα παιδιά, περνάει από ελέγχους έτσι ώστε να είναι ασφαλές ε, για τη χρήση του, στη χρήση του από το παιδί. Αυτό δεν ισχύει πάντα για τις συσκευές, ε, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες προς το χρήση, χρήστη. Και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συνέπειες. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που θα σας παρουσιάσει ορισμένες άλλες πτυχές του ζητήματος. Ευχαριστώ, Φερνάντο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω διαφορές εθνικών νομοθεσιών. Λοιπόν, μια διαρκής πρόκληση στον μέτρη της εργασίας κατά του κυβερνού εγκλήματος. Τα σημερινά εργαλεία δεν υπαρκούν για το έγκλημα του αύριο. Οι εγκληματίες εξελίσσονται, εμείς παρακολουθούμε σχετικά αργά. Τόσο αφορά τους ε, ουσιώδες ε, κανόνες όσο και τους δικονομικούς κανόνες. Ε, το θέμα της ε, δικαιοδοσίας, το θέμα της ε, ετεροδικίας κλπ. Έχουμε διαφορετικές νομικές παραδόσεις επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον ρόλο της αστυνομία, των εισαγγελέων, τη συλλογή και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων κλπ. Δεν υπάρχει λοιπόν εναρμονισμένο πλαίσιο για τις σχετικές έρευνες, τις μυστικές έρευνες, ιδιαίτερα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Όσον αφορά την ε, διεθνή συνεργασία, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία στην αμοιβαία αρρώγη. Εδώ προχωρήσαμε αργά, δεν εξυπηρετούμε τις επιχειρησιακές ανάγκες. Τα κείμενα που έχουν ε, συγγραφεί και ψηφιστεί δεν έχουν γραφτεί με το διαδίκτυο στο μυαλό. Αν και στην οδηγία υπάρχουν συγκεκριμένα όρια όσον αφορά την, το παραδεκτό των τεκμηρίων, πρέπει να σημειωθεί πολύ μεγαλύτερη πρόοδος. Αυτή τη στιγμή μόνο λίγα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία η οποία θα σε ισχύ σε έναν μήνα από σήμερα. Η τελευταία κατηγορία αφορά την ταχύα εξέλιξη της τεχνολογίας. Ακόμα και οι ειδικοί δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ των μη ειδικών και της τεχνολογίας ο στόχος μας παραμένει βεβαίως, να μπορούμε να προσεγάγουμε τους υπευθύνου. χρειάζεται ελάχιστη τεχνογνωσία, εννοείται, πρέπει να εκπαιδευτούν και οι εισαγγελείς, οι δικαστές, χρειαζόμαστε καλύτερη και περισσότερη λοιπόν εκπαίδευση. Επόμενη διαφάνεια. Το διαδίκτυο μας διευκολύνει, αλλά είναι και τεράστιο εμπόδιο. Μας επιτρέπει να επικοινωνούμε, να καταναλώνουμε, να ψυχούμεθα, να επιχειρούμε να κάνουμε δουλειές, όμως επιτρέπει και στο έγκλημα να ανθεί και πολλές φορές δυσκολεύει τις απαγγελίες κατηγοριών. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση. Και εδώ όμως ήμασταν αργοί. Χρειάζονται λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Εδώ τονίζω ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Για να βρούμε λύσεις πρέπει να επιτύχουμε έναν επαρκή συγκερασμό μεταξύ των δικαιωμάτων αφενός και, των, και της δράσης της αστυνομία, των εισαγγελέων κλπ. Η εφαρμογή όλων αυτών πρέπει να συνάδει με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα και θυμίζω βέβαια ότι όπως πάντα ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Δεν έχω λοιπόν κάποιε έτοιμε λύσει, μαγικές λύσει σήμερα, απλώ σχολιάζω τον μηχανισμό που χρησιμοποιεί σήμερα η Europol για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει στο πεδίο καθημερινά. Προ τούτο χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία. Επόμενη διαφάνεια, καινοτομούμε λοιπόν, μελετούμε το έγκλημα όσο πιο καλά μπορούμε, πίσω από κάποια επιτυχημένη έρευνα, υπάρχει επαρκής έρευνα. Οι σημερινοί τρόποι, όπως είπα, δεν επαρκούν. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από κάθε εγκληματική δραστηριότητα, το χρήμα και ούτω καθεξής. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι οι οργανώσεις αυτές στον κυβερνοχώρο δεν είναι παραδοσιακές. Δεν υπάρχει παραδοσιακή ιεραρχία. Πολλές φορές ε, συστήνονται και διαλύονται εντάχει ε, και σε αυτά ακριβώ τα χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμοστούμε. Το νομικό μας πλαίσιο, παραλαμβάνω, δεν είναι προσαρμοσμένο. Πρέπει να ενημερωθεί, αλλά να μην ξεχνούμε την νομολογία η οποία θα αξιοποιηθεί για να ενισχύσουμε το πλωστάσιό μας κατά του εγκλήματος. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε μέχρι να βρούμε τις τελικές λύσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να επαγγέλουμε κατηγορίες, να προσάγουμε και χρειαζόμαστε και εναλλακτικέ λύσεις ε, όσον αφορά την αμοιβαία αρρωγή. Χρειάζεται οι δικαστικέ αρχέ να εμπλέκονται από νωρί, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και τη διεθνή συνεργασία. Και χρειαζόμαστε δίκτυα, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη, πλατφόρμες και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράσει στην πράξη για να αντιμετωπίσουμε, να καταπολεμήσουμε με τρόπο αξιόπιστο το νέο έγκλημα. Το EUCDF, το οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Europol και η Eurojust είναι ένα εργαλείο. Εγκατακλείδη λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτές με καινοτομία, με συνεργασία και με συνεργασία στην καινοτομία. Με αυτά κλείνω και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Άλλους δύο μιλητές έχουμε και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Γκράχαμ Βίλμοντ, ε, τμήματάρχη ε, αρμόδιο για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το μοιραστούμε λίγο με τον συνάδελφο από την Προστασία των Δεδομένων, τμήματάρχης, ε, και εκείνος για να σας δείξουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προελίσσαντες ομιλητές έθεσαν το πλαίσιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και οι απαντήσεις που θα δώσουμε μπορούν να εγγραφούν σε 4-5 τίτλους. Ποιο είναι το κεκτημένο όταν μιλούμε για νέες πολιτικές για τις ε, δίωξη του εγκλήματος. Το δεύτερο φορά την απάτη. Θα μιλήσω για τη σύμβαση Βουδαπέστη Βουδαπέστης του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης και τέσσερα, ε, για τη στρατηγική μας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αρχίζω από το κεκτημένο. Υπάρχει οδηγία του 2013 για τις επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικά. Βλέπουμε πώς τα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία και πώς την εφαρμόζουν και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους για να ε, βελτιωθεί η εφαρμογή της οδηγίας και αν χρειαστεί να αναλάβουμε και δράση ε, επί παραλήψη. Τι κάνει λοιπόν αυτή η οδηγία, να αρμονίζει ε, τον ορισμό της επίθεσης κατά πληροφοριακών συστημάτων και εναρμονίζει ε, τα, ε, τις ποινικέ κυρώσεις. Και ορίζει επίσης και τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Ε, προχωρώ στις ε, εξελίξεις ε, της πολιτικής δίωξη του εγκλήματος. Αυτή είναι η βασική μας αποστολή όταν έχει ένταλμα η αστυνομία να αποκομίσει ε, αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ δεν πρόκειται για μαζική παρακολούθηση του πληθυσμού. Έχουμε εξαιρετική αγαστή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη και άλλες γενικές διευθύνσει και οργανισμούς τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Europol και η Eurojust εδώ παρόντε. Αυτό που μας ενδιαφέρει, υπάρχουν ε, στοιχεία πρώτον μπορεί οι ιδιοκτικέ αρχές να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ε, στοιχεία, μπορούν να τα διαβάσουν, είναι κρυπτογραφημένα. Ε, για την αποθήκευση ή την ε, παρακράτηση στοιχείων υπάρχει μια δικαστική απόφαση του Δεκεμβρίου και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλες συζητήσεις για το κατά πόσο μπορούν οι διοκτικές αρχές να διατηρούν, να αποθηκεύουν αυτά τα στοιχεία. Το Συμβούλιο και η Προεδρία έχει στήσει μια ομάδα εργασία για να τα κοιτάξει αυτά τα θέματα και από την επιχειρησιακή σκοπιά και από την νομική. Και η πρώτη ε, συνεδρίαση ασχολήθηκε και αυτή η ομάδα των φίλων της Προεδρίας ε, έχει ακόμα πολλή δουλειά για τα επόμενα τις επόμενες συνεδριάσεις, αυτό βέβαια δεν είναι δικό μου θέμα. Επίσης, θα πρέπει εμεί να βοηθούμε τα κράτη-μέλη ε, με κάποια καθοδήγηση για το πώς να ευθυγραμμίσουν την νομοθεσία τους για να την κάνουν συμβατή με την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό χρειάζεται μελέτη, λεπτομερή και προσεκτική και της απόφασης και του ε, κάστοτε εθνικού ε, νομικού πλαισίου και της ομάδας των φίλων της Προεδρίας προχωρώ στα ηλεκτρονικά στοιχεία και πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ τον κύριο Μάκνομ για τα καλά του λόγια. Και πάλι εδώ έχουμε μια τρεπλή προσέγγιση. Πρώτον, θέλουμε να ε, βελτιώσουμε την άμεση συνεργασία των διοκτικών αρχών των κρατών μελών με τους παρόχους υπηρεσιών ε, διαδικτύου. Επίσης, ε, θέλουμε να βελτιωθεί ε, το σύστημα συνεργασίας και αμοιβαία δικαστικής συνδρομής με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αντίστοιχα εντάλματα και τις εντολές. Ε, στη συνέχεια, το τρίτο, να ζητούμε κοινέ λύσεις για την επιβολή ε, του νόμου σε μια δικαιοδοσία, τι γίνεται με τις διασυνοριακές περιπτώσεις και πώς τα κράτη-μέλη τις αντιμετωπίζουν η διαδικασία είναι χωρίς αποκλεισμούς, όπως σας είπα, ε, συνεργαζόμαστε με τις διοκτικές αρχές των κρατών μελών, τα Υπουργεία, τους οργανισμούς Eurojust Europol και ε, βεβαίως με τους ενδιαφερομένους στον κλάδο της οικονομίας αυτό. Πολύ σημαντικό. Θα προτείνουμε μια δέσμη μέτρων και εναλλακτικών τον Ιούνιο και θα επανέλθουμε σε λίγους μήνες, σε δύο μήνες από τώρα, για να σας ε, πούμε πιο ουσιαστικά. Το τελικό στοιχείο διαδικασία κρυπτογράφησης είναι πιο πρόσφατη. Μόλις αρχές του έτους ε, άρχισε να μας απασχολεί. Εδώ πρόκειται για μια διαδικασία σε δύο στάδια. Πρώτα χρειάζεται συλλογή των πληροφοριών και αυτή τη στιγμή έχουμε όλες τις πληροφορίες από όλους τους ενδιαφερομένους να τις αναλύσουμε και πάλι να ε, προτείνουμε μια δέσμη μέτρων. Πρώτον, με ποιους συνομιλούμε τώρα, σε ποιους απευθυνόμαστε εδώ. Η βασική ενεχόμενη είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, Europol, Eurojust, η ΕΝΙΣΑ για τα θέματα της ασφάλειας του διαδικτύου και ε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θέλω να τονίσω εδώ το ρόλο του έχουν κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι μόνο φιλοσοφικές αναζητήσεις και αγωνίες, αλλά πολύ συγκεκριμένα αυτά που προτείνουν. Ε, τους επόμενους δύο μήνες θα ζητήσουμε από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να διοργανώσουν εργαστήρια, συζητήσεις με πυρογνώμονες των, των μελών ε, σε δύο παράλληλες διαδικασίες, μια τεχνική και μια νομοθετική νομική πώς συνδέεται με την τεχνολογία του διαδικτύου, είναι το ένα το τεχνικό σκέλος και το νομικό σκέλος είναι ε, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη που διέπουν ε, τη χρήση τέτοιων τεχνικών από τις διοκτικές αρχές για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και πώς όλα αυτά εγγράφονται στα πλαίσια των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για μας είναι σημαντικό να μην ανάγεται η συζήτηση μόνο να περιορίζεται στον ευάλωτο χαρακτήρα κάποιων στοιχείων. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά υπάρχουν και άλλα και τεχνικά και νομικά που πρέπει να ε, μελετήσουμε πάρα πολύ. Βεβαίω έχουμε σχέδια για ε, πρόταση νομοθεσία, αλλά ε, αφήνουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για να τα αναλύσουμε, να μελετήσουμε και να δικαιολογήσουμε τι θα προτείνουμε ή τι δεν θα προτείνουμε στο τέλος της διαδικασίας. Ε, πρόθεσή μας είναι να κάνουμε την τελική πρόταση τον Οκτώβριο. Όλα αυτά τα θέματα ε, θέτουν ε, ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οπότε θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το θέμα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και, τα, ε, η προστασία τους, ε, γιατί μιλάμε για ένα θεμελιώδες δικαιωμά, είναι ύψης της σημασίας. Και θα πρέπει να πληρούνται οι προαπαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν θέλουμε ε, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχει επιγραμμική ασφάλεια αλλά και ιδιωτικότητα από την άλλη. Το ε, ένα δεν, αποκλείει το, δεν πρέπει να αποκλείει το άλλο, αλλά να αλληλοϊποστηρίζονται. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε και τις κατάλληλες τεχνικές και νομικές λύσεις για την ε, προστασία τους όταν μιλάμε για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ε, διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία για εγκληματικές δραστηριότητες θα πρέπει να σεβαστούμε το πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων και εάν υπάρχει παρέμβαση ε, στο θέμα της προστασίας, αυτός ο παρεμβατισμός θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι δικλείδες ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή πέρυσι μάλλον εγκρίναμε την ε, προστασία προσωπικών δεδομένων, τον κανονισμό για την ε, προστασία προσωπικών δεδομένων θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου του 2018 και ορισμένα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για τη σημερινή συζήτηση. Το GDPR και πώς τα στοιχεία ενός παρόχου και η μεταβίβαση αυτή οριοθετείται. Και αυτό σημαίνει ότι η αποκάλυψη στοιχείων από τους παρόχους στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βασίζεται σε μία από τις έξι ε, βασικές, ε, βασικά άρθρα του GDPR. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να δούμε τι ισχύει στην οδηγία 9546 μέσα στα πλαίσια της νόμιμης ε, αποκάλυψης και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα για εμπορικούς σκοπούς και για την πρόληψη του εγκλήματος. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα ισχύει με βάση νομοθετικά δεδομένα. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων μας δίνει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τη μεταβίβαση προσωπικών ε, δεδομένων ενός παρόχου σε μία τρίτη χώρα. Αυτά είναι παραδείγματα περιπτώσεων όπου ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας δίνει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κύβερνο χώρο. Επίσης υπάρχει και ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων από πλευράς συνεργασίας αστυνομικών και δικαιοδοτικών αρχών θα ισχύσει από το 2018 για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Να υπάρχει δηλαδή καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, των διοκτικών αρχών μάλλον των κρατών μελών και να οικοδομηθεί και ένα κλίμα εμπιστοσύνη σε σχέση με την νομική ασφάλεια. Η οδηγία όταν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε μια καλύτερη συνεργασία καταπολέμησης του εγκλήματος. Στο μέλλον χρειάζεται να ανταλλάσσουμε ένα και περισσότερες πληροφορίες και φυσικά και με οργανισμούς όπως η Europol και η Eurojust και αυτή η οδηγία ορίζει ένα κοινό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Η οδηγία αυτή δεν αφορά περιορισμό της εφαρμογής του νόμου, αλλά στην, αφορά τη σωστή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι στα πλαίσια καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το αίτημα των διοκτικών αρχών στον πάροχο ζητά προσωπικά στοιχεία, ας πούμε διεύθυνση IP. Γι' αυτό η οδηγία αυτή θέτει τους όρους επεξεργασίας δεδομένου και ιδιαίτερα το άρθρο 39 της οδηγίας ε, σε σχέση με τους παρόχους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Τελευταία. Πρόθεση να κλείσουμε. Α, συγγνώμη. Νομίζω ότι είχαμε 15 λεπτά ως Κομισιόν, αλλά τα τρία τελευταία σημεία που θέλω να θίξουμε πολύ περίπτυχα είναι. Βλέπουμε ταχύτατη ανάπτυξη της ε, απάτης στον των νομισμάτων. Υπάρχει η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά τις πλαστικές κάρτες. Έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για μια πιθανή πρωτοβουλία. Θα έχουμε και μια μελέτη επιπτώσεων. Θα συζητήσουμε αυτό το Σεπτέμβριο. Δύο πράγματα ακόμη. Έχουμε επίση τη Σύμβαση τη Βουδαπέστη, του Συμβουλίου τη Ευρώπη που διέπει τις περισσότερες δραστηριότητες μας στον τομέα αυτών. Υποστηρίζουμε πλήρως την σύμβαση αυτή και συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα σε τρίτες χώρες. Τέλος, όσον αφορά τη στρατηγική για την ασφάλεια στον χώρο ως το 2013, και την αναθεώρησή της. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να την αναθεωρήσουμε και θα προβούμε σε αξιολόγηση και θα λάβουμε και τις σχετικές αποφάσεις, πιθανότερα εντός των προσεχών εβδομάδων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την υπομονή σας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για όλες τις εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω στην, την προσοχή σας στο ότι έχουμε εδώ ένα έντυπο το οποίο μπορείτε να πάρετε μαζί σας μετά το πέρας της συζητήσεως. Και τώρα, ο λόγος στην κυρία Ελίσσα Βόζεμπεργκ από το ΕΛΚ ε, ως εισηγητρία. Πρόεδρε, ε, καταρχάς ε, έχω οριστεί ραπορτέρ για το, την, για το report σχετικά με το έγκλημα στο διαδίκτυο Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές σήμερα για τις εξαιρετικά εξειδικευμένες αν και σύντομες λόγω του χρόνου εισηγήσει για τα επιμέρους θέματα που κάθε ένας εξ αυτών ε, έχει επεξεργαστεί. Να πούμε ότι η κοινή παραδοχή όλων μας είναι ότι το έγκλημα στο διαδίκτυο, οι εγκληματίες και η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις διοκτικές αρχές και κυρίως από την νομοθεσία μας. Αυτό συμβαίνει διότι εκ των πραγμάτων, πέραν των άλλων στοιχείων, η νομοθεσία για την εναρμόνισή της είτε στον τομέα της πρόληψης είτε στον τομέα της καταστολής θέλει μια γενικότερη ευρωπαϊκή αντίληψη η οποία όπως πολύ σωστά επισημάνα το καθένας μέσα από την ειδικότητά του δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ε, εστιάζω σε ένα μείζον πρόβλημα το γεγονός ότι δεν έχουμε μία εναρμονισμένη νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη σαν μια νομοθεσία ομπρέλα που να υπερβαίνει την, τον χαρακτήρα των επιμέρους οδηγιών για επιμέρους ζητήματα έτσι ώστε να μπορούμε είτε στον τομέα της πρόληψης είτε στον τομέα της καταστολής να γίνουμε αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα, επειδή αυτό το οποίο λέω μπορεί να είναι πολύπλοκο, άλλωστε πολύπλοκη είναι όλη η διαδικασία της έρευνας, όπως έχετε επισημάνει και του τρόπου της ανακάλυψης, πρόληψης αφενός καταστολής αφετέρου του εγκλήματος μέσα στο, στον κυβερνοχώρο, ένα εξειδικευμένο θέμα για το οποίο ε, θα υποβάλω και την ερώτησή μου, είναι ε, παραδείγματος χάρη τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Ξέρετε ότι θα μπορούσε ας πούμε η συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε, σε επίπεδο νομοθεσίας να προσκρούει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος να διαφέρει ο τρόπος της φύλαξης των ιχνών, ο τρόπος της ε, διατήρησης ε, δικαιώματος χρήσης και ε, δικαιώματο χρήση πέραν από το κράτο μέλο και σε άλλα κράτη-μέλη των προσωπικών δεδομένων. Ο τρόπο που κάθε κράτο μέλο, καλυπτόμενο, ε, δεν το λέω αρνητικά, πίσω από την επικουρικότητα, έχει μια νομοθεσία η οποία δεν είναι συμβατή προ άλλα κράτη-μέλη πόσο μάλλον και από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα λοιπόν, αφού ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τι πολύ εμπεριστατωμένε εισηγήσει, να ρωτήσω πόσο υπάρχει στη σκέψη της Επιτροπής εν ώψη των παρατηρήσεων του Ιουνίου οι νομοθετικέ πρωτοβουλίε εναρμόνισης της νομοθεσίας για τον τρόπο χρήση των ηλεκτρονικών ε, και ιχνών και κυρίω των αποδεικτικών μέσων. Ε, με μόνο να σκεφτεί κανείς αν υπάρχει μια συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ηλεκτρονικών σε τέτοιο εξελιγμένο επίπεδο ώστε να εξαρθρωθεί μια εγκληματική οργάνωση σε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν επιτρέπει τη χρήση αυτών των στοιχείων, η υπόθεση όλη έχει καταρρεύσει. Με αυτό το σκεπτικό και πάλι σας ευχαριστώ και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Okay, thank you. Uh, I would like Ευχαριστώ. Κυρία Μύρια Μντάλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν σήμερα στην Επιτροπή μας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και πιστεύω ότι αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι ε, συνεχώς αλλάζει το κυβερνό έγκλημα. Κάποιος είπε ότι είναι πολύ μπροστά οι εγκληματίες και εμείς ολιγορούμε. Θα, για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε έτσι με κριτικό μάτι τα εργαλεία και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, τις ελλείψεις, τις αδυναμίες, να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και οι σημερινές και οι Η οδηγία μας το 2013 κατά ε, ε, των επιθέσεων σε πληροφορικά συστήματα χρειάζεται ε, αναβάθμιση, χρειάζεται βελτίωση. Ας πούμε, ε, το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος σήμερα. Βέβαια δεν αρκεί μόνο να προσαρμόσουμε την οδηγία αυτή, θα πρέπει ε, να αξιολογήσουμε την πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών στο διαδίκτυο. Εγώ είμαι εισηγήτρια από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε για αυτό το θέμα. Και ορισμένοι εμπειρογνώμονε αναφέρθηκαν ε, επανελειμμένα στο γεγονό ότι η καταπολέμηση του ηλεκτρονικό εγκλήματος δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διακυβεύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών μας. Και επιχαίρομαι για την οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτική ζωή και την προστασία της και το Κοινοβούλιο ελπίζω να ε, εγκρίνει την πρόταση που θα φέρει η διαπραγματευτική ομάδα. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Κάποια στιγμή στην αρχή αρχή της ακρόασης ακούσαμε για τα θέματα της ε, ετεροδικίας και τα θέματα ε, της εδαφικής επικράτησης ενός κράτους μέλους. Θα είπε ο κύριος Δελασαπέλ, που μπορεί να είναι εμπόδιο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτά τα πράγματα δεν γνωρίζουν σύνορα, ούτε υπήρους, ούτε περιφέρειες. Δεν αρκεί λοιπόν να εξετάζουμε το θέμα μόνο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που υπερβαίνει τα σύνορά μας. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, αν δεν απατώμε, το είπε ο κύριος Φερνάντο Ρουίθ, όταν μίλησε για την ασφάλεια των συσκευών. Αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, δεν θα έρθουμε πάλι αντιμέτωποι με τις διαφορές, της δικαιοδοσίες ε, στην ένωμη τάξη των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε κατευθύνσεις γραμμές. Πώς μπορούμε αυτό να το εναρμονίσουμε δεν έχει να κάνει μόνο με τον ευάλωτο χαρακτήρα και το πόσο μπορούμε να είμαστε θύματα μιας κατάστασης. Είναι και ευκαιρίες αυτές που ανοίγονται. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς ο κόσμος θα αντιμετωπίζει και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών ε, στο διαδίκτυο. Πρόσφατα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι γίνεται διαφήμιση ε, στους νέους hacker για να ε, αξιοποιήσουμε τις δεξιότητές τους. Βέβαια, σε βαθμό που είναι νόμιμα αυτά, ε, υπάρχουν καριέρες έτσι σταδιοδρομίες που ανοίγονται ελπιδοφόρες και κερδοφόρες. κάτι άλλο που άκουσα είναι ότι οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες ε, θέλουν να προσλαμβάνουν hackers γιατί υπάρχουν τα bounties, είναι κάποια συστήματα που πρέπει να χακάρουν οι hackers έτσι ώστε να μην τους χακάρουν τους ίδιους κάποιοι άλλοι κακόβουλοι. Ε, με χαρά θα συνεργαστώ με τους άλλους κυριοσυγητές και ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ναταλή Κρισπέκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για αυτή την ε, παρουσίαση, αυτές τις διασταυρούμενες παρουσιάσεις τεχνικής υφής. Τώρα έχουμε καθυστερήσει, γι' αυτό δεν θα επεκταθώ, αλλά αφού διαβάσω την παρουσίασή τους θα σας υποβάλω ερωτήσεις ε, γραπτός για, για αυτή τη θεματική που έχει μεγάλη σημασία και μας απασχόλησε και στην προηγούμενη ως προς την προηγούμενη έκθεση που έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Στο ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχουν αυτές οι απειλές, ο πολλαπλωσιασμός τους και οι διαφορετικές πηγές των απειλών που χρήζουν απάντησης δεν θα ήθελα να προβάλλω αντιρρήσεις αποκλειστικά εμείς είμαστε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν είμαστε πολύ άριθμοι εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε επί νομοθετικών κειμένων. Μιλήσαμε για ε, κείμενα και ιδιαίτερα την οδηγία του 2013. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο, κατά την άποψή σας, χρειαζόμαστε πραγματικά μια νέα νομοθεσία και μιλώ για ένα αριθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε νέα μέσα ή αυτά που προϋπάρχουν αρκούν. Γιατί αναλωνόμαστε σε θέματα, επιμέρους θέματα και ούτω καθεξής. Μιλάμε για περισσότερη εναρμόνιση, συνεργασία αλλά κυνηγάμε την ουρά μας στην ουσία ενδεχομένως. Εάν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με διάφορες ε, τεχνικές ε, αντιμετώπισης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτό το άοσμο υλικό υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές στον χώρο. Δεν έχουμε λοιπόν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης. Χρειάζεται να νομοθετήσουμε εκ νέου και αν ναι, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεύτερον, ε, σαν συνέχεια της πρώτης ερώτησης, στην Λίλη, στη χώρα μου, έγινε ένα φόρουμ αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στις αρχές του 2017 και φαίνεται ότι το ποινικό οπλοστάσιο καταπολέμησης του εγκλήματος του κυβερνοχώρου προϋπάρχει, μπορεί να είναι διάσπαρτο, αλλά προϋπάρχει. Άρα δεν χρειαζόμαστε νέα νομοθετικά μέσα, αλλά χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους. Άρα, ρωτώ, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη κατάρτισης των δικαστών σε αυτό το τομέα. Πρόκειται για πρόσφατα γεγονότα. Επίσης, το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο, σήμερα το πρωί διάβασα στον τύπο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να γνωμοδοτήσει εκ νέου στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής ευρωπαϊκής ατζέντας. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Είμαι σκιώδης και γι' αυτό μακρηγορώ ή θέλω απαντήσεις. Ε, κύριε Πρόεδρε, μπορούν οι ομιλητές να μου στείλουν και γραπτώσεις απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα ε, δεν θα μπορούσε να προωθήσει το θέμα, να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με τη συζήτηση με τον Επίτροπο Τζούλιαν Κίνγκ, Μιλήσαμε για θέματα ανθεκτικότητας, δηλαδή μιλάμε για έναν προληπτικό άξονα ή έχετε περαιτέρω στοιχεία ε, έτσι ώστε να μπορέσετε να διελευκάνετε το ζήτημα. Μίλησα για τρία το πολύ τέσσερα λεπτά. Okay, thank you very much. Ε, ε, then... Οπότε, να συνεχίσουμε με απαντήσει ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την περίφημη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ εσάς και τους βουλευτές που έθεσαν ερωτήματα. Ρωτήσετε, θα καταθέσουμε νομοθετικές προτάσεις. Αυτό ακριβώ σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα στοιχεία ιδιαίτερα, τα τεκμήρια. Και τον Ιούνιο, όπως είπα, θα παρέλθουμε με σειρά εναλλακτικών προτάσεων και θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι όριμες νομοθετικές προτάσεις ή κάποια βάση απλώς συζήτησης. Αυτό ακριβώς εξετάζουμε αυτήν τη στιγμή. Επίσης μας ρωτήσετε μήπως κυνηγάμε την ουρά μας κλπ. Ε, αρκεί να ενισχύσουμε τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Το δεν αποκλείει το άλλο. Αυτή είναι η απάντησή μας. Είτε καταθέσουμε νομοθετικές προτάσεις, σίγουρα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων, την παροχή επιπλέον εκπαίδευσης. Θα δούμε αν χρειαζόμαστε μεγαλύτερα οικονομικά μέσα, υπολογιστέ, ανθρώπους κλπ. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε σε όλους τους τομείς δηλαδή που προανέφερα. Ρωτήσετε επίσης τι γίνεται με τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων και τη σχετική οδηγία και τι γίνεται με την ασφάλεια του διαδικτύου των πραγμάτων του Internet of Things και τι γίνεται με τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής που ελέγχουν ψηφορίες τα εξετάζουμε αυτά στο πλαίσιο τη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Θα δούμε αν χρειαζόμαστε αναθεώρηση αυτή τη στρατηγική. Η Κομισιόν λοιπόν αυτή τη στιγμή μελετά ενδελεχώ όλα τα σχετικά θέματα και θα απαντήσει με τρόπο ολοκληρωμένο όσον αφορά το σύνολο τη στρατηγική ή κάποια τμήματά τη. Επίση, αναφερθήκατε στο τμήμα εκμετάλλευση των παιδιών ασχολούμαι με αυτό. Ε, δεν είχα έρθει προετοιμασμένο, Αύριο ο υποδιευθυντή μα θα σα μιλήσει από ό,τι ξέρω, οπότε δεν υπάρχει λόγο να αναφερθώ σήμερα στο ζήτημα γιατί θα το καλύψει αύριο τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, παιδιών. Όσον αφορά τώρα την ενδιάμεση αναθεώρηση τη νομοθεσία για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Δυστυχώ δεν έχουμε μαζί μα συναδέλφου που γνωρίζουν το θέμα, αλλά ξέρω ότι εργάζονται εντατικά. Αν θέλετε, ευχαρίστω να μεταφέρω το ερώτημα στου αρμοδίου συναδέλφου. Καμία αντίρρηση. Τέλος. Η αντοχή και η ενίσχυση της αντοχής των συστημάτων μας είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε στο πλαίσιο της ενδεχόμενης ε, αναθεώρησης της στρατηγικής μας για τον κυβερνοχώρο και το διαδικτύο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπερτράν Σαπέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σύντομα να απαντήσω σε κάποια σχόλια και ερωτήσεις που έγιναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ το θέμα των ορισμών και των λέξεων. Η εναρμόνιση ε, και η συνεργασία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ έχουμε πρόβλημα να εναρμονίσουμε στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μία από τις έννοιες που έχει αναδειθεί είναι η νομική διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, ε, με τις δικονομικές εγγυήσεις και διεπιφάνειες μεταξύ ε, των φορέων ε, διασυνοριακά και όχι εναρμόνιση αυτή καθ' αυτή. Αντίστοιχα, αν θέλουμε να έχουμε νέα εργαλεία, γίνεται μια ερώτηση, χρειάζονται νέα μέσα και νέα εργαλεία. Το νέο έχει να κάνει με νέα κείμενα ε, στην κείμενη νομοθεσία. Μπορεί να χρειάζονται νέα μέσα διεθνούς συνεργασίας που μπορεί να μην είναι νομοθεσία, μπορεί να μην είναι συμβάσεις και συνθήκες, αλλά κάτι ε, άλλο που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε στάνταρ και πρότυπα πολιτικής που χρησιμοποιούν ε, οι εταίροι που συνεργάζονται ε, σε επίπεδο υπηρεσιών ή σε επίπεδο νομικών κειμένων. Η νομική λοιπόν διαλειτουργικότητα, legal interoperability και policy standards. Και κάτι άλλο που έχει να κάνει με την κλίμακα ε, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι ενέφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαν ότι έχει τη μοναδική ευκαιρία τώρα να ε, ηγηθεί και να δημιουργήσει πρότυπα. Ταυτόχρονα όμως τα πρότυπα αυτά ε, πολιτικής και η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να έχουν και μία κλίμακα σε μεγαλύτερες περιφέρειες. Εκεί που δρούν οι φορείς, δηλαδή πώς μεταφέρεις σε μία μεγαλύτερη κλίμακα ε, ε, αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να διαφεύγουν όσο γίνεται λιγότερη παράδειση εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και επίσης ε, το θέμα της δικαιοδοσίας είναι κάτι το οποίο αφορά πολλούς τομείς και όχι μόνο το δικό μας και αυτό που διακυβεύεται κυρίως είναι πώς ασκεί κανείς κυριαρχία στην ψηφιακή εποχή. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Ήταν εξαντλητική και εκτενέστατη. Ε, σας ευχαριστώ που συνοψίσατε για τις παρατηρήσεις, για τις ε, παρεμβάσεις σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και σας θυμίζω ότι υπάρχει και η μελέτη αυτή, μερικά αντίτυπα στην είσοδο της αίθουσας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9, καλό σας βράδυ.